So, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, μια και δεν έχει έρθει ο πρόεδρος της Επιτροπής, μου ζητήθηκε να προεδρεύσω. Δεν ξέρω όμως γιατί, διότι είμαι πρεσβύτερος εδώ. Άραγε. Ε, το αφήνω στη δική σας κρίση, γιατί ε, μου ζήτησαν να προεδρεύσω. Ελπίζω πάντως ότι η πρόεδρός μας θα θα έρθει, αλλά είναι μία... είναι τιμή για μένα και ευχαρίστησή μου να καλωσορίσω τον ομιλητή μας σήμερα, τον Αχμέτ Μπιν Μοχάμεντ Αλ Τζαρβουάν, τον πρόεδρο του Αραβικού Κοινοβουλίου. Σας, ε, θα θέλω να σας καλωσορίσω και σας ε, εξοχότατε και τον πρέσβη. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να μας δώσετε ό,τι πληροφορίες ε, χρειάζεστε, θέλετε μάλλον, και μετά θα ακούσουμε και τους συναδέλφους και μόλις έρθει η πρόεδρος θα αποχωρήσω διακριτικά. Εξοχότατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, γιατί θα είναι πιο εύκολο για μένα να μιλήσω αραβικά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα ε, που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να συναντήσω μαζί με τους συναδέλφους μου την Επιτροπή σας μέσα στα πλαίσια της ε, συνεργασίας ανάμεσα στα δύο κοινοβούλια. Ελπίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια και θα ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στα δύο κοινοβούλια μας. Ελπίζουμε ότι η σημερινή συνεδρίαση θα είναι το πρώτο βήμα ε, για να υπάρξει μια συνεργασία σε πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί φιλίας που ενώνουν τους λαούς μας. Αυτή την περίοδο εμείς στις αραβικές χώρες προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποιους ε, δημοκρατικούς θεσμούς μεταξύ αυτών και το Αραβικό Κοινοβούλιο και θέλουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις με διεθνή όργανο όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με τα ε, περιφερειακά ή εθνικά κοινοβούλια η, Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ε, συνδέεται με τον αραβικό κόσμο και μέσω των οικονομικών συμφερόντων αλλά και μέσω δεσμών οφειλίας. Έχουν ε, συναυθεί συμφωνίες συνεργασίας ε, ανάμεσα στον αραβικό κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η τάση αν θέλετε έχει υλοποιηθεί με την υπογραφή συμφωνιών με διάφορες αραβικές χώρες και υπάρχει και μία υπογραφή συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών σαν ε, συνέχεια της ε, διαδικασίας της Βαρκελόνης και της ε, Ένωσης για την Μεσόγειο αλλά και την συνεργασία με τις χώρες του κόλπου μετά την ε, συμφωνία που υπογράφηκε το 1989. Εμείς ε, σαν εκπρόσωποι των λαών μας ε, δεν, δεν πρέπει να αρκούμεθα μόνο σε μια παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω, να ενισχύσουμε την συνεργασία μέσω διμερών συμφωνιών. Και Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις προτάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, όσον αφορά τον αραβικό κόσμο και την κατάσταση στην ε, Μέση Ανατολή, το, την, τις Ισραηλινο-Παλαιστινιακές διαφορές και θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κοινοί στόχοι, κοινά συμφέροντα ανάμεσά μας και ελπίζουμε ότι θα ε, ενισχύσουμε τις κοινέ αρχές και τα ιδανικά ε, για την ειρήνη κυρίως, τις ανθρώπινες αξίες, τα κοινωνικά κεκτημένα, ε, εμείς ε, απορρίπτουμε ε, κάθε διαφορετική αντιμετώπιση των λαών με βάση την γλώσσα ή τη θρησκεία. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λαοί έχουν κάθε δικαίωμα να επιλέξουν την, την πορεία τους χωρίς να να υπάρχει οποιαδήποτε ανάμιξη από το εξωτερικό. Ε, πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να ε, χειραγωγούμε τους λαούς ε, ή τις χώρες, κυρίως στην Μέση Ανατολή θα πρέπει να προωθήσουμε κάποιες πολιτικές αφοπλισμού και θα πρέπει να προωθήσουμε την ειρήνη. Βέβαια υποστηρίζουμε τις κοινέ αξίες, τα κοινά συμφέροντα που ενώνουν τους θεσμούς, τους δικούς σας και τους, δικός, τους δικούς μας. Τώρα όσον αφορά την Συρία, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τον αραβικό κόσμο αλλά και από, την, ε, και από τους δυτικούς ε, για να ε, δημιουργηθεί μια κυβέρνηση δημοκρατική και για να περιορίσουμε τον ε, Άσαντ βλέπουμε ότι ε, υπάρχει μία σύγκρουση ανάμεσα στις αρχές στους, στους εξωτερικούς στους από το εξωτερικό και αυτοί που το πληρώνουν είναι ο λαός της Συρίας. Βλέπουμε ότι ένοπλες ομάδες διαπράττουν δολοφονίες καθημερινά ε, βλέπουμε τον αριθμό των προσφύγων ο οποίος ε, εκτοξεύεται. Ε, δεν έχουμε λύσεις στην διάθεσή μας και δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θέλουν δυστυχώς να, συνεχίσει, να, συνεχίσουν, να συνεχίσει σύραξη για να ικανοποιήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Άρα θα πρέπει όλοι να είμαστε προσακτικοί έτσι ώστε τέτοιου είδους συγκρούσεις να μην διαιωνιστούν διότι ε, απλώς και μόνο αποσταθεροποιείται η περιοχή, δεν εξυπηρετείται το συμφέρον κανενός, καμιάς χώρας και... Ε, αποσταθεροποιούνται και οι σχέσεις με του εταίρου μας, τους Ευρωπαίους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να δοθεί ένα τέλος ε, σε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει όλοι όσοι διαπράττουν ε, δολοφονίες ε, να σταματήσουν Βέβαια είναι σίγουρο ότι θα, υπάρξει μια πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος έτσι ώστε να, σταματήσουν, να σταματήσει η ένοπλη σύγκρουση και να βρεθεί μια δημοκρατική λύση η οποία να δώσει μια απάντηση στις δημοκρατικές ε, επιθυμίες του Συριακού λαού θα πρέπει και να ικανοποιηθεί και το αίτημα των Συρίων να ε, υπάρξει ένα πολυκομματικό σύστημα και στη χώρα τους. Θα πρέπει ε, να δοθεί, ε, θέλετε, ένα σαφές μήνυμα και προς τον Συριακό λαό ότι τον υποστηρίζουμε. Θα ήθελα να σας πω ότι έχει διευρυνθεί ούτως ή άλλως ο τομέας συνεργασίας ανάμεσά μας σε πολλούς τομείς, στον οικονομικό, στον ε, κοινωνικό τομέα. Υπάρχει η Μεσόγειος, το Μάρεν Nostrum, που αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον, στην ευρωπαϊκή κοινωνία και στην αραβική κοινωνία, που ε, το μόνο που ζητάνε είναι να συνυπάρχουν ειρηνικά. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις και ελπίζουμε ότι θα έχετε ε, και εσείς μια σαφή θέση, μια σαφή στάση όσον αφορά στις ε, παρεμβα... εξωτερικές παρεμβάσεις στον αραβικό κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή που δώσατε στα... στο μήνυμά μου και ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Επιτροπής και ελπίζω ότι οι εργασίες μας θα είναι ε, καρποφόρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και για αυτή την εισαγωγή που και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο Τένοκ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν ανέμενα να μιλήσω πρώτο. Είναι μεγάλη τιμή για την ομάδα μου να έχουμε τον πρώτο αγορητή. Καλώ ήρθατε κύριε Πρόεδρε του Αραβικού Κοινοβουλίου. Είμαι ένα από του ιδρυτέ ε, των φίλων ε, τη ε, ομάδα συνεργασία με τι χώρε του κόλπου και έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τι χώρε τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και την Αραβική Άνοιξη και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Και πιστεύω ακράδαντα, όντα στο Ευρωκοινοβούλιο για 14 χρόνια, ότι μια κοινοβουλευτική συνιστόσα είναι ιδιαίτερα σημαντική σε όλα τα εκτελεστικά πολιτικά σώματα. Του δίνει μεγαλύτερη νομιμότητα και διασφαλίζει και μια λογοδοσία ή εξέταση των πραγμάτων από τα όσα τεκταίνονται. Και ιδιαίτερα σημειώνουμε το ε, ενδιαφέρον και την αύξηση σε σχέση με τον Αραβικό Σύνδεσμο με ρόλο κλειδί που είχε στην παρέμβαση στη Λιβύη για παράδειγμα να απαλλαγεί αυτή η χώρα από το δικτάτορα Καντάφη που την ταλάνιζε και πιστεύω απόλυτα ότι το Αραβικό Κοινοβούλιο θα συνεισφέρει σε αυτή την κοινοβουλευτική συνιστόσα στη διαμόρφωση των πραγμάτων στον Αραβικό κόσμο αλλά και παγκόσμια. Και αυτό το Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο παραδοσιακά έχει και ισχυρούς δεσμούς με άλλα υπερ εθνικά σώματα. Είμαι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας αυτού του Ευρωκοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και αναμένουμε ότι θα υπάρξει και μια αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης διότι θα ε, ενταχθεί στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ε, το Ευρωκοινοβούλιο. Και καθώς ομιλούμε σήμερα και χθε υπήρχε μεγάλη συνάντηση του Ευρωδικτύου Euronet των ε, χωρών της Ανατολικής Συνιστώσας και οι Αρμένοι συνάδελφοι για πρώτη φορά είναι ενδιαφέρον ότι συνήλθαν μαζί μας και είχαμε και έναν διάλογο μαζί τους ε, και αυτό διανοίγει δυνατότητες μεταξύ χωρών που πολλές φορές βρίσκονται σε εχθρικές σχέσεις μεταξύ τους όπως οι Αρμένοι με τους Αζέρους. Ε, ένα τέτοιο φόρουμ δίνει μια ευκαιρία επαφών και η Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση ασυνήθιση σε αυτές τις διαστάσεις που έδωσε την δυνατότητα ε, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι από τις χώρες της Αφρικής και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Ισραήλ να μπορέσουν να συνέλθουν και να συζητήσουν για την προαγωγή της ειρηνευτικής διεργασίας στη Μέση Ανατολή. Και στην Αιθιοπία πέσει είδαμε πάλι ότι το Ευρωκοινοβούλιο που υποστηρίζει ιδιαίτερα και οικονομικά και με συμβουλευτική συνδρομή στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και την Αφρικανική Ένωση. Πολλά περισσότερα θα μπορούσαν να γίνουν λοιπόν για την ε, διασταυρούμενη, διασταυρούμενη αυτή γονιμοποίηση μεταξύ των κοινοβουλίων μας είναι νομίζω το μεγαλύτερο υπερεθνικό άμεσα ε, εκλεγμένο από τους πολίτες ε, κοινοβουλευτικό σώμα παγκόσμια και είμαι υπερήφανος πανικός σε αυτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ακόμα και όντας Βρετανός Ευρωβουλευτής βέβαια σε παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής ε, και σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε ε, στις αρχές ε, πριν από λίγο δηλαδή την ενδέκατη επέτειο της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας σε σχέση με την αραβική αυτή πρωτοβουλία και υπάρχει κάποια δυνατότητα να επανενεργοποιηθεί αυτό το θνησιγενές εγχείρημα και την δυνατότητα οι Ηνωμένε Πολιτείε να συνεισφέρουν στην ειρηνευτική διαδικασία. Είναι αυτή η προφανή επιλογή η Αραβική Πρωτοβουλία για την Ειρήνη. Και είναι ενδιαφέρον και η, ενδιαφέρουσα η απόφαση, επίμαχη βέβαια, για την άρση του εμπάργου όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του καθεστώτος της Συρίας. Η χώρα μου, Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία ανέλαβαν ρόλο πρωτοπόρων γι' αυτό, επειδή είχε διχαστεί η Ευρώπη. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να είναι θετικό και να διασφαλίσουμε ότι οι μετριοπαθείς αντάρτες θα πάρουν αυτά τα όπλα και δεν θα διοχετευτούν αλλού αυτά τα όπλα και για την Γενέβη 2 υπό τις διεργασίες αυτές θα μπορούσαν με τη στήριξη των ΗΠΑ και των Ρώσων να προλιάνουν το έδαφος για μια αλλαγή καθεστοτική στη Συρία και ένα άλλο θέμα το οποίο και αυτό βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο δεν συζητήθηκε χθε, αλλά θα συζητηθεί άμεσα η Χεσμολά και το στρατιωτικό σκέλος να εγγραφεί τις τρομοκρατικές οργανώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε και μια επίθεση στη Βουλγαρία κατά Ισραηλινών τουριστών και έχουμε και μια αντίστοιχη επίθεση και στην Κύπρο που κρύβεται πίσω από αυτά τα γεγονότα η Χεσμολά και ίσως αλλάζουν και άποψη και οι Γάλλοι. Ίσως θα θέλατε να σχολιάσετε το γεγονός μια και είναι μέρος της κυβέρνησης στο Λίβανο και σε σχέση με το δικό σας κοινοβούλιο πώς θα μπορούσε αυτό να συνεισφέρει στην σταθεροποίηση της κατάστασης αν για παράδειγμα αυτοί ε, αποτελέσουν τμήμα αυτού του καταλόγου τρομοκρατικών οργανώσεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Τένοκ, λέει ο Πρόεδρο. Η απαγόρευση εξαγωγής όπλων ε, δεν ε, ήρθε αλλά δεν παρατάθηκε. Στο αποτέλεσμα όμω είναι το αποτέλεσμα το ίδιο. Η κυρία Νέτς παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε του Αραβικού Κοινοβουλίου, Μιας και είχαμε την ευκαιρία προηγουμένως να μιλήσουμε λιγάκι στα γαλλικά κατεδία, να μιλήσω κι εγώ έρχομαι την άδειά σας, να σας ευχηθώ το καλώς ήρθατε εξ ονόματος του Κοινοβουλίου μας και της δική μου πολιτική πολιτικής ομάδας των φιλελευθέρων. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Εδώ και κάποιους μήνες, κύριε Πρόεδρε, διερωτώ με όλο και περισσότερο για το εξή. Ο Αραβικός Σύνδεσμος, η διάσκεψη των Ισλαμικών χωρών, το Συμβούλιο Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου. Όλοι αυτοί οι φορείς που είναι διακρατικοί όπου συμμετέχουν μέλη κυβερνήσεων και κοινοβουλίων των αραβικών χωρών ή μουσουλμανικών χωρών. Και καταλαβαίνω απολύτω ότι δεν είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα, δεν είναι ταυτόσιμε οι έννοιε, δεν τα συγχαίω. Αλλά συναντώνται συχνά. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν από αυτό το πρίσμα να πάρουν θέση ως προς την σύγκρουση Σουνιτών και Σιητών. Αυτό που πραγματικά διχάζει και καθιστά ανέφικτη την δημιουργία μιας αραβικής ε, ολοκλήρωσης που καθίσταται έτσι αδύνατη. Βλέπετε να υπάρχει η πιθανότητα να αναπτυχθεί κάποια πρωτοβουλία, κάποια δράση, ώστε να γίνουν ε, λιγότερο βίες αυτές οι συγκρούσεις και ενδεχομένως να βρεθεί κάποια διέξοδος, διότι μου φαίνεται αναντήρητο, και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση από αυτού, μου φαίνεται αναντήρητο λοιπόν ότι περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα του πληθυσμού παγκοσμίω οι ίδιες οι μουσουλμανικές ομάδες, οι ομάδες των μουσουλμάνων πολιτών είναι θύματα αυτών των συγκρούσεων. Αυτοί χάνουν τη ζωή τους κατά δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. <clears throat> Αυτή είναι η ερώτησή μου. Θα θέλαμε πολύ να βοηθήσουμε. Αλλά εμείς δεν είμαστε οι πλέον αρμόδιοι για να απαντήσουμε σε τέτοιο ζήτημα. Θα μπορούσατε εσείς να μας πείτε κάτι. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμερ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσυπογράψω σε όσα πάνε συνάδελφοι. Για τη σημασία που αποδίδει το Ευρωκοινοβούλιο στην δράση μπορεί να αναλάβει το δικό σας κοινοβούλιο, διαρθρώνοντας την δράση διαφορετικών φορέων. Υπ' αυτήν την έννοια, να ρωτήσω το εξής. Ε, ζήτημα που είναι πολύ σχετικό με το ρόλο που έχετε αναλάβει. Μάλιστα. Την περασμένη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο κιόλα. Μπερδεύτηκα ήδη. Ξεκίνησε η εξέταση της έκθεση από το Freedom House για την ελευθερία των μέσων επικοινωνία ε, στον κόσμο και την έκφραση, την ελευθερία της έκφραση ε, στον κόσμο. Κάποιε χώρε τα πήγαν πολύ καλά, είχαν καλή βαθμολογία σε αυτήν την αξιολόγηση. Και βεβαίως τα ελεύθερα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι θεμελιώδους σημασία στοιχείο για τη λογοδοσία των κοινοβουλίων βεβαίως, εφόσον τα κοινοβούλια θέλουν να έχουν κάποια παρακολούθηση και κάποια εποπτεία του θέματος. Τι πιστεύετε εσείς ότι το δικό σας κοινοβούλιο θα μπορούσε να κάνει ως προς αυτό το σκοπό. Ένας άλλος τομέας που μας ενδιέφερε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, για τον οποίο μάλιστα πρόσφατα εγκρίναμε την περασμένη εβδομάδα κιόλα ένα ψήφισμα, είναι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Εδώ ε, εντοπίσαμε τις ευθύνες μας το να βοηθήσουμε τις χώρες της Ελλαδικής Άνοιξης να ε, ανακτήσουν περιουσιακά του στοιχεία που είχαν ε, καταχραστεί τα προηγούμενα δικτατορικά καθεστώτα. Πολλά από αυτά είναι παγωμένα σε δικές μας χώρες, στη δική μας επικράτεια, αλλά πολλά βρίσκονται και στις δικές σας χώρες, συγκεκριμένα στις χώρες του κόλπου. Τι πρωτοβουλίε λοιπόν ο Αραβικό Σύνδεσμο και πιο συγκεκριμένα το Αραβικό Κοινοβούλιο μπορούν να αναλάβουν για να ενισχύσουν τι προσπάθειε των χωρών που επιδιώκουν κάτι τέτοιο. Είναι θέμα αξιοπρέπεια. Είναι θέμα οικονομική ανάγκη επίση για πολλέ από αυτέ. Και είναι και θέμα δικαιοσύνη. Θα χρειαστούν όποια βοήθεια τους μπορεί να τους προσφερθεί. Τι βλέπουμε όμως. Μια άλλη παρενέργεια είναι η κουβετιανή εταιρεία η οποία κέρδισε πρόσφατα μια δίκη, μάλλον μια περίπτωση διαιτησίας για τη Λιβύ, από τη Λιβύη, την κέρδισε τη Λιβύη στο δικαστήριο, από κέρδη που δεν αποκομίστηκαν από ένα σχέδιο αναπτυξιακό που είχε κανονίσει ο Καντάφη με αυτή την κουβεθιανή ε, εταιρεία. Είναι μια άλλη οπτική γωνία, στρεβλή του ίδιου προβλήματος όμως. Και το ανέφερε και ο συνάδελφος, ο κύριος Τάνο, και εδώ θέλω να έρθω στη δεύτερη παρατήρησή μου. Η αραβική πρωτοβουλία, πού είναι, πού πηγαίνει για τη Συρία. Πηγαίνει κάπου ή δεν πηγαίνει πουθενά. Είχαμε προηγουμένως τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα. Μας είπε ότι το ζήτημα της Συρίας θα προκαλέσει μια άλλη περίπτωση σαν το Αφγανιστάν στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε η σύραξη στη Συρία να εξελίσσεται σε πόλεμο που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας. Περιφερειακές διαστάσεις λαμβάνει και μάλιστα κοντεύει να γίνει πόλεμος μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας ή των Σιητών και των Σουνιτών. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας ευχαριστήσω όλους και όλες για τις ερωτήσεις σας, που ήταν όλες πολύ έκστοχες, διότι πραγματικά τέτοιου είδου διάλογος είναι το θεμέλιο της σχέσης συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων μας. Ελπίζω να υπάρχει πραγματικά μια καλύτερη και σχέση μεταξύ των κοινοβουλίων μας, ώστε να βρούμε λύσεις ή να καταλήξουμε σε αποτελέσματα τα οποία να είναι επωφελή και για τις δύο πλευρές απαντώντας ε, στην ερώτηση για την ειρηνευτική διαδικασία στην ε, Μέση Ανατολή. Στον αραβικό κόσμο έχουμε επανειλημμένως εκφραστεί υπέρ της ειρήνης. Θέλουμε την ειρήνη. Η θρησκεία μας, οι παραδόσεις μας βασίζονται στην ειρήνη. Την ειρήνη στα πλαίσια της θρησκείας. Πάντοτε στηρίζαμε οποιαδήποτε ηγεσία του αραβικού κόσμου που προσανατολιζόταν προς την διευθέτηση του, προβλέ... του προβλήματος της ε, σύγκρουσης Ισραηλινών Αράβων. Θέλαμε λοιπόν μια πρωτοβουλία που να συγκλίνει σε αυτό το στόχο και πιστεύουμε ότι είναι νόμιμα τα δικαιώματα που προβάλλει ο Παλαιστινιακός λαός να ζει σε ένα δικό του κράτος, ένα κράτος ασφαλές, με ασφαλή σύνορα και θα πρέπει να βοηθηθεί. Ως προς την ειρηνευτική λοιπόν διαδικασία την στηρίζουμε. Εάν το Αραβικό Κοινοβούλιο κληθεί να παραστεί στις ε, διαπραγματεύσεις, ευχαρίστως να συμμετάσχουμε και να στηρίξουμε αυτήν την πορεία. Σε ό,τι αφορά τα όπλα ή την άρση του εμπάργου για την πώληση όπλων στην περίπτωση της Συρίας, δεν θέλουμε να υποδαβλήσουμε τα πάθη εδώ. Δεν θέλουμε να υπάρξει εξοπλισμός μαζικής καταστροφής και να φτάσει ως τη Συρία. Ε, το καθεστώς, το επίσημο καθεστώς της Συρίας διαπράττει δολοφονίες, σκοτώνει νέους, παιδιά, λιγότερο νέους, άμαχους. Αυτό το καταδικάζει το κοινοβουλίο μας. Είμαστε κατά του πολέμου. Θέλουμε μία λύση ειρηνική και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι προσπάθειες γίνονται, αλλά θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις, χρειάζονται δράσεις εδώ, πράξεις. Εδώ και δύο χρόνια, δύο χρόνια είναι σε εμφύλιο πόλεμο η Συρία. Μέχρι πού θα φτάσει αυτό. Πού θα φτάσει αυτός ο πόλεμος, οι διαφορετικές εντμαχόμενες πλευρές και οι εξωτερικοί παρατηρητές παίζουν πολύ περίπου διαφορετικούς ρόλους, ακόμη και στο, στο πλαίσιο του αραβικού κόσμου. Βεβαίω, η οπτική γωνία των Ευρωπαίων διαφέρει πολύ από αυτή των Αράβων, αλλά ουσιαστικά οδηγούμαστε σε αστάθεια ολόκληρη τη περιφέρεια αυτή, τη γεωγραφική περιοχή. Δεν ωφελεί αυτό τα κοινά μα συμφέροντα, γιατί είμαστε υπέρ τη διεθνού ειρήνη, όπω είπα, τη παγκόσμια ειρήνη. Ο πόλεμο λοιπόν στη Συρία πρέπει να πάυσει, διότι οι βιοπραγίε, οι τρομοκρατικέ ενέργειε μπορεί να εκπορευθούν από αυτή την κατάσταση. Στηρίζουμε λοιπόν οποιονδήποτε, οποιοδήποτε φορέα ή πλευρά ε, προδοθεί μια λύση του ζητήματος της Συρίας. Λύση που βέβαια καλό θα ήταν να βρεθεί εκ των έσω, αλλά εξωτερικοί συμμετέχοντες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη, το Ευρωκοινοβούλιο, πρέπει να διαδραματίσουν ένα ρόλο καθοριστικό και ή δυνατόν θετικό πρόσφορο για την εξέβρεση μιας λύσης. Είπαμε ότι θα οργανώσουμε συναντήσεις, συνομιλίες, περιμέναμε τη δεύτερη θητεία του κυρίου Ομπάμα, την επανεκλογή του. Περιμένουμε πάρα πολύ. Καθυστερούμε. Η ανάληψη καθηκόντων από τον κύριο Ομπάμα για δεύτερη φορά δεν έδωσε ακόμα κανένα ευεργετικό αποτέλεσμα. Τι θα κάνουμε τώρα, θα περιμένουμε να αλλάξει πρόεδρο και το Ιράν προκειμένου να εξετάσουμε με προσοχή αυτό το θέμα, υπό διαφορετική οπτική γωνία, δεν είναι λύση αυτό. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά των όπλων που χρησιμοποιεί το, η κυβέρνηση, που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις του Ασάντ. Μιλάμε για όπλα ρωσικής και ιρανικής προέλευσης. Εδώ λοιπόν καταδικάζουμε ως εκπρόσωποι του αραβικού κόσμου όλη αυτή την ε, εξέλιξη. Σε ό,τι φορά τη Χεσμολά, και εδώ θα απαντήσω σε παρατηρήσεις και ερωτήσεις που έγιναν. Στον αραβικό κόσμο και ιδίως στο αραβικό κοινοβούλιο είμαστε μουσουλμανικής ε, θρησκείας, Σουνίτες, Ιήτες, Δρούζοι, Χριστιανοί. Όλοι βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή και κάτω από την αιγίδα του αραβικού κόσμου. Δεν θέλουμε να έρχονται εξωτερικοί φορεί και να ρίχνουν λάδι στη φωτιά στον αραβικό κόσμο. Δεν θέλουμε καμία παρέμβαση, είτε του Ιράν, είτε τη Ευρώπη, είτε των Πολιτειών. Όλοι αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε βία η σύγκρουση και σε διάσπαση του αραβικού κόσμου. Αυτό το καταδικάζουμε. Σε ό,τι αφορά τη Χεσμολάχ, το Αραβικό Κοινοβούλιο πριν από ένα τρίμηνο κιόλα δήλωσε ότι η εξακολούθηση του πολέμου στη Συρία μπορεί να προκαλέσει την ανάμειξη και άλλων εξωτερικών φορέων. Ο, το, Λίβανος έχει πληγεί ήδη από τον πόλεμο αυτό και αυτό είναι μόνο η αρχή. Είναι μια χώρα που είναι προσφυλή στον αραβικό κόσμο ο Λιβανός. Είναι μια χώρα επίσης που την αγαπούν ιδιαίτερα και οι Ευρωπαίοι. Δεν θέλουμε το Ιράκ να συμπαρασυρθεί από την κρίση στη Συρία. Δεν θέλουμε ούτε η Ορδανία να συμπαρασυρθεί Μιλάμε για χώρε που είναι όμορε τη Συρία, αραβικέ χώρε. Και εμεί ω εκπρόσωποι των αραβικών λαών καλούμε εδώ. Απευθύνουμε έκκληση στην, από το βήμα αυτό, το λαμπρό αυτό βήμα, τε, απευθύνουμε έκκληση να ενώσετε τις φωνές μας σας με τις δικές μας ώστε να αναζητήσουμε λύσεις σε διεθνές επίπεδο προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ να λάβουν αποφάσεις για να δοθεί ένα τέρμα σε αυτή την σφαγή στη Συρία, να ξεκινήσει ένας πραγματικός διάλογος, να σταματήσει η μηχανή του πολέμου. Πράγμα που δεν θα γίνει αν δεν αρχίσει διάλογος για τη Συρία και για τα θέματα της Συρίας. Σε ό,τι αφορά τις κοινέ μας εργασίες. Ήρθαμε από τις διάφορες αραβικές χώρες, χώρες που μεταξύ τους είναι εταίροι και μας ενώνουν με την Ευρώπη βεβαίως, σχέσεις ε, παλιές που πάνε πολύ μακριά στο παρελθόν. Αυτές τις σχέσεις θέλουμε να τις διατηρήσουμε, να τις ενισχύσουμε και να τις καλλιεργήσουμε. Οι πολίτες λοιπόν της Ευρώπης και οι δικοί μας προς όφελος των μελλοντικών γενεών, προς όφελος των Αράβων που κατοικούν στην Ευρώπη, πρέπει να ασχοληθούν με τις πολιτικές, τις πολιτιστικές, τις εμπορικές μας σχέσεις. Αυτές θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με τους φίλους και φίλες βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου και θέλουμε να δημιουργηθεί μια κοινή μεθοδολογία, ένας κοινό μηχανισμός συνεργασίας, μια κοινή ομάδα, μια κοινή επιτροπή που να επιτρέπει την ενίσχυση της συνεργασίας, των σχέσεων συνεργασίας να επιδιώκει την προάσπιση των αραβικών συμφερόντων ε, στην Ευρώπη και την προάσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων στις αραβικές χώρες. Μας ενδιαφέρει να συγκεντρώσουμε πληροφορίες στο σωστό πλαίσιο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάποιες φορές ε, επιμένουν σε μία οπτική γωνία και παραμελούν μια άλλη. Το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο μπορούν εδώ να διδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, ώστε να διοχετεύουν τις ορθές πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που ανέφερε η κυρία Γκόμες, υπάρχουν τέτοια περιουσιακά στοιχεία, υπάρχει περιουσία, περιουσία ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και αυτά ακόμη βρίσκονται στα χέρια των ε, εκτότων καθεστώτων. Το Αραβικό Κοινοβούλιο για την ώρα δεν έχει λάβει κανένα αίτημα να εξετάσει κάποιο τέτοιο θέμα. Στις αρχές των κοινοβουλευτικών μας εργασιών επικεντρωθήκαμε σε υποθέσεις που αφορούσαν όλες τις αραβικές χώρες. Συγκεντρωθήκαμε στα στοιχεία που μας ενώνουν και αφήσαμε κατά μέρος αυτά που μας χωρίζουν. Επικεντρωθήκαμε και εξετάσαμε ποια, ποιοι παράγοντες ενισχύουν τις σχέσεις μας με την Ευρώπη, με την Ασία και το επαναλαμβάνω εδώ. Δεν θα θέλαμε καμία διαταραχή στις σχέσεις μας. Δεν θέλουμε να θέσουμε ερωτήσεις που φέρνουν κάποιον σε δυσάρεστη θέση ή που μπορεί να αντίκενται στα συμφέροντα των εταίρων μας. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας, με εσάς και την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ προκειμένου να ε, στρέψουμε το βλέμμα προς τους ορίζοντες συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα όσα μας είπατε κύριε Πρόεδρε και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι μαζί σας ως ένα πολυμερές κοινοβούλιο μπορούμε, θα έπρεπε να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε τη σχέση μας ε, και να περάσουμε σε, σε βάθος συζητήσεις, ε, να συζητήσουμε για τη σύραξη στην Μέση Ανατολή η τετραμερίσα ε, και ο Αραβικός Σύνδεσμος θα έπρεπε να συνεργαστούν στενότερα σε αυτό το πλαίσιο και σίγουρα είναι και το θέμα των κοινοβουλευτικών διάβλων σημαντική υπόθεση που θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτό και να μπορέσουμε να ασκήσουμε την επιρροή μας στα τεκτενόμενα ώστε η φωνή μας αυτή, το μέσο αυτό να ενδυναμωθεί. Και καταστήσατε σαφές σε σχέση με την σύραξη στη Συρία πόσο πρέπει να είναι δική μας υπόθεση να μην υπάρξει αποσταθεροποίηση με την ανάμειξη άλλων χωρών, όπως τώρα για παράδειγμα συμβαίνει στο Λίβανο ή ε, στο, στην Ιορδανία και να μπορέσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει για να αποφύγουμε μια τέτοια αποσταθεροποίηση. Όμως, καταδεικνύεται ότι τέτοιες κρίσεις σήμερα δεν μπορούν αυτόματα να θεωρηθούν ότι σταματούν στα σύνορα μιας χώρης, χώρας. Έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις και γι' αυτόν τον λόγο χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας με αυτή την ευκαιρία σήμερα και με τις επαφές που είχατε και με τον πρόεδρο Σούλτς θα μπορέσουμε να διευρύνουμε αυτές τις σχέσεις και επαφές μας ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε την επιρροή μας που πρέπει και το οφείλουμε στους πολίτες μας να το κάνουμε ώστε η κοινοβουλευτική μας επιρροή ως επίδραση να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτό το κοινοβουλευτικό πλαίσιο εξέφρασα την ικανοποίησή μου για το ότι κατά το πρώτο ήμιση της θητείας σας ε, εξελέγητε κατά το 2012 αν τα θυμάμαι σωστά ήρθατε σε εμάς στις Βρυξέλλες ε, και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα με τους συναδέλφους σας που είναι εδώ παρόντες και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του δικού σας Κοινοβουλίου σε αντιπροσωπεία που βρίσκονται οι συνάδελφοι εδώ να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις και να βρούμε τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε αυτό το πλαίσιο επαφών. Σας ευχαριστώ που ήρθατε.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

στο κανάλι. και und Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να χαιρετήσω ανάμεσά μας Χαιρετήσω τον κύριο Κόμπλερ ανάμεσά μας, ειδικό εντεταλμένο, απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση στο Ιράκ. Σας ευχαριστούμε θερμά που εκ νέου ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο σε εμά. Γνωρίζουμε με ποιες δυσκολίες παλεύει το Ιράκ και επίσης με ποιες δυσκολίες και εσείς ο ίδιος παλεύετε προσωπικά και πρέπει ρητά να εκφράσω και να πω ότι έχω ιδιαίτερη εκτίμηση για το έργο των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράκ και για την προσωπική σας δουλειά και εμπλοκή εκεί. Πώς τα τελευταία δύο χρόνια έχετε συνεισφέρει με το έργο σας στο Ιράκ η εντολή σας νομίζω εκπνέει και θα λάβετε νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα και θα ήθελα να πω για τέτοιες προϋποθέσεις, υπό τέτοιες προϋποθέσεις να συνεχίζετε το έργο δεν είναι το ευκολότερο και θα μπορούσε κανεί να το πει αυτό για τις ευθύνε σας. Ο Απρίλιος ήταν ο πιο θανατηφόρος μήνας των τελευταίων ετών στις αντιπαραθέσεις σειράξεις μεταξύ Σουνιτών και Σιητών των δύο αυτών κοινοτήτων που οξύνονται οι αντιπαραθέσεις σειράξεις τους. 700 νεκροί, 700 θάνατοι κατά τον μήνα Απρίλιο, άμαχοι περισσότεροι. Και υπάρχουν και διασυνδέσεις ή επαφές και με την βία που από την ίδια τη Συρία περνά και εκρήγνεται στο Ιράκ η κατάσταση στα Ιρακινο-Συριακά σύνορα και στην δυτική περιοχή του Άνμπαρ δεν διευκολύνει καθόλου τα πράγματα. Και θα έλεγα και ότι από δικής μας πλευράς εμείς, σε σχέση με τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες και την, τον ρόλο τους στο Ιράκ, θα πρέπει να συνεισφέρουν ώστε να τερματιστεί η βία και να μπορέσει το Ιράκ να ειρηνεύσει. Νομίζω είναι μια εξέλιξη που πρέπει να αναχαιτήσουμε αυτή, αυτή της ε, έκριθμης βίας με τα τόσα πολλά θύματα τα οποία προκάλεσε τα τελευταία χρόνια. Κύριε Κόμπλερ, έχετε λοιπόν τον λόγο παρακαλώ. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και θα περάσω στην επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Εθνών και θα σας προσφωνήσω στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά που είμαι ενώπιον σας. Ήμουνα εδώ πριν από ένα έτος και έχω την τιμή να σας προσφωνήσω. Πολλά πράγματα συνέβησαν αυτό το τελευταίο έτος. Και όπως εσείς αναφέρατε ο ίδιος στην εισαγωγή σας, η Ιρακινή, το Ιράκ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή και ανησυχώ ιδιαίτερα. Ανησυχώ ιδιαίτερα επειδή η χώρα πραγματικά βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και υπάρχει κίνδυνος να οπισθοδρομήσει προς τους κινδύνους του παρελθόντος 2006-2007 είχα γνωρίσει την κατάσταση και ήμουν πρέσβης στο Ιράκ της Γερμανίας και κανείς δεν θέλει να ξαναζήσει αυτές τις φρικαλές περιόδους εμφυλίου πολέμου με σειράξεις όλων εναντίον όλων. Δεν θέλουμε να πιστοχωρήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Η κλιμακούμενη βία μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Πέθαναν, σκοτώθηκαν 85 ε, προχθές, ε, εχθές 27. Είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει άμεσα και όπως είπατε εσείς Πρόεδρε είναι πολύ σημαντικό να απευθύνουμε έκκληση στους πολιτικούς, διότι είναι δική τους ευθύνη να σταματήσουν την αιματοχυσία σε αυτή τη χώρα. Και αυτό θα έπρεπε να γίνει όχι μόνο από εμά, αλλά και από τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Λόγοι Λόγοι είναι τα ανεπίλητα προβλήματα στο Ιράκ. Έχουμε ένα, μια διακούσα κατάσταση, λιμνάζουσα κατάσταση από το 2010 με, μετά τη συμφωνία του Αρμπίλ που ποτέ δεν εφαρμόστηκε και την αυξανόμενη απογοήτευση και απόγνωση των Σουνιτών και την αντίδρασή τους να κατεβαίνουν στους δρόμους και να διαδηλώνουν από πέρσι το Δεκέμβριο. Πέρσι το Δεκέμβριο που μετά από την ε, ε, δολοφονία ε, και τις διαδηλώσεις που είχαν καταλήξει στους δρόμους οι περισσότερες ήταν ειρηνικές στους δρόμους του Ανμπάρ της Νινεβή και πάρα πολλοί Σουνίτες που ζουν εκεί όλοι τώρα φοβούνται ότι αυτό το φάσμα το φάσμα του εμφύλιου πολέμου θα επανέλθει, θα επιστρέψει στο Ιράκ. Ένας άλλος ε, παράγοντας κλιμακούμενης βίας, οξυνόμενο πρόβλημα, είναι η βία στη Συρία και οι επιπτώσεις. Θα μπορούσε κανείς ε, να δώσει μια περίληψη λέγοντας συγχώνευση ε, σειράξεων. Και όλοι βλέπουμε ότι ανησυχούν με την ε, Συρία, εξετάζουμε οι περισσότεροι το Ιράκ, όμως η διεθνής κοινότητα δεν κάνει λόγο για το Ιράκ, διότι επικεντρώνεται στη Συρία. Όμως συγχωνεύονται τα πεδία μαχών και φυσικά η Συρία έχει επιπτώσεις στους Σουνίτες του Ιράκ, η κατάσταση στη Συρία. Φυσικά έχουν κάποια αιτήματα ε, εκείνοι που κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις. Εμείς από τα Ηνωμένα Έθνη δεν είμαστε υπέρ του ενός ή του άλλου. Πρέπει η συνταγματική διαδικασία να ακολουθηθεί για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα πολιτικών αιτημάτων τα περισσότερα αιτήματα των διαδηλωτών που οδηγούν και σε βία αυτές οι διαδηλώσεις αφορούν την πολιτική δομή του Ιράκ. Υπάρχουν πολλά όχι. Όχι στην ενότητα του Ιράκ. Ναι, υπέ της απόσχησης περιφερειών και περιοχών. Το θέμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου τα νομοθετήματα για την αμνίστευση. Όλα αυτά είναι πολιτικά αιτήματα και ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη σοβαρά από την κυβέρνηση. Τώρα υπάρχει μια αφωνία, αφασία μεταξύ των κομμάτων. Δεν επικοινωνούν, δεν συζητούν τα κόμματα μεταξύ τους, δεν συνέρχονται, δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχει ημερήσια διάταξη, ατζέντα για ένα τέτοιο διάλογο. Και αυτό οδήγησε αυτή τη χώρα στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Τι κάνουμε τώρα εμείς ως Ηνωμένα Έθνη και τι θα μπορούσε να πράξει η διεθνής κοινότητα. Αυτό που κάναμε από τον Ιανουάριο πέρυσι, όταν η κατάσταση ουσιαστικά επιδεινώθηκε με τις διαδηλώσεις και που οδήγησαν επίσης ε, και στα ε, ε, συμβάντα της Χαμπίτζα όπου 42-43 άτομα δολοφονήθηκαν σε μια πλατεία όπου διαδήλωναν και αυτό ήταν πώς να το πω, ένα σοβαρότατο προηγούμενο, ένα σοβαρότατο συμβάν σε σχέση με την σχέση των διαδηλωτών και της κυβέρνησης. Αυτό που κάνουμε τι είναι. Κρατάμε ίσες αποστάσεις και από τις δύο πλευρές και από την, με την κυβέρνηση με την οποία έχουμε επαφές και σχέσεις αλλά έχουμε αποστάσεις, ίσες αποστάσεις και με τους διαδηλωτές. Δεν τοποθετούμαστε επί των πολιτικών τους αιτημάτων αλλά επικεντρωνόμαστε στο αίτημα για διάλογο. Προσπαθούμε να συνέρθουμε με όλους τους είτε στο Ιράκ στο Ραμάντι Πάμε στο Ραμάντι. Είμαστε οι μόνοι διεθνεί εκπρόσωποι που πάμε στο Ραμάντι, στη Σαμάρα, στη Φαλούτζα, στην Τικρίτ, σε όλε αυτέ τι περιοχέ όπου βρίσκονται διαδηλωτέ Σουνίτε. Αλλά επίση και στο ε, Αρμπίλ, στο Αμάν, στο ε, Ντουμπάι, όπου η αντίσταση των Σουνιτών ε, έχει έδρα και δραστηριοποιούνται. Προσπαθούμε να του οδηγήσουμε γύρω από ένα τραπέζι για διάλογο και ειρήνη και ειρήνευση λέγοντας ότι δεν συμμετέχουμε παίρνοντας ε, μέρος υπέρ του ενός ή του άλλου και προσπαθούμε να έχουμε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους ε, στα πολιτικά αιτήματα, έχουμε πέντε αρχές επί των οποίων ε, βασίζουμε το έργο μας. Και η πρώτη αρχή είναι το να διατηρηθεί η ενότητα της χώρας και η ακαιρεότητα της χώρας γεωγραφικά και οποιοδήποτε θέλει να διαλύσει αυτή τη χώρα, να υπάρξει κάποια απόσχηση περιοχής, τουλάχιστον σε πολιτικά αιτήματα, είμαστε ε, κάθετα εναντίον. Πρώτον λοιπόν διασφάλιση ενότητας του Ιράκ. Δεύτερη αρχή, η αρχή της μη άσκησης βίας. Όλοι πραγματικά φοβούνται ότι η τάση επανέρχεται να ασκείται βία, να έχουμε πολιτοφυλακές, να έχουμε θανάτους αμάχων. Η αρχή λοιπόν της μη άσκησης βίας. Τρίτη αρχή, η μη σεκταριανή ε, πορεία. Είναι σημαντικό να δει κανείς ότι όλο και πιο ακραία γίνεται η γλώσσα. Οι ε, ακραίες θρησκευτικές τάσεις και τοποθετήσεις είναι κάτι που και από τις δύο πλευρές πρέπει να υπάρξει έργο και από τους θρησκευτικούς ηγέτες και από τους ίδιους τους διαδηλωτές να μειωθεί αυτό το εύρος. Ιδιαίτερα η ρητορική ε, των ακραίων. Δεν πρέπει να ξαναγυρίσει αυτή η χώρα στην αντιπαράθεση Σιητών, Σουνιτών όπως στο παρελθόν. Η τέταρτη αρχή υπέρ τη οποία είμαστε είναι ότι όλες οι συζητήσεις θα πρέπει να διεξάγονται επί τη βάση του συντάγματο. Αυτό είναι το ανώτατο νομοθέτημα της χώρας. Είναι ο μόνος νόμος που έχουν οι πολίτες, το σύνταγμα του Ιράκ. Βλέπουμε λοιπόν στις συζητήσει μας με τους διαδηλωτέ ε, των Σουνιτών που οδηγούν σε αυτές τις βιοπραγίε ένα όλο και μεγαλύτερο όχι. Όχι στο Σύνταγμα, όχι στον Πρωθυπουργό. Θέλουμε αυτό να το μεταμορφώσουμε σε μια πολιτική του ναι, καταφατική, υπέρ του Συντάγματος, υπέρ της πολιτικής ε, ομαλότητας. Δεν είναι τέλειο το Σύνταγμα, δεν υλοποιείται για παράδειγμα. Το Ιράκ είναι μια ομοσπονδιακή χώρα, όμως ο ομοσπονδιακός αυτός χαρακτήρας δεν τον παίρνουν στα σοβαρά στο Ιράκ. Δεν υπάρχει στην πρακτική εφαρμογή άσκηση αυτής της ομοσπονδιακής αρχής. Όμως δεν είναι δυνατόν να πόσχει κανείς από το Σύνταγμα, να παρεκκλίνει από το Σύνταγμα και από την ένωμη τάξη. Η συνέπεια θα είναι στο μέλλον ότι θα πρέπει στο, με, το Σύνταγμα να μπορέσουν να προχωρήσουν και ομοσπονδιακός χαρακτήρας τι σημαίνει να μπορούν να έχουν εξουσίες οι επαρχίες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει δεύτερο σώμα, δεν υπάρχει ε, συμβούλιο των ε, επαρχιών, δεν, δεν μπορεί να λειτουργήσει ομοσπονδιακός αυτός χαρακτήρας χωρίς στο δεύτερο κοινοβουλευτικό σώμα. Και το πιο σημαντικό φυσικά είναι το θέμα και τη ε, της συμμετοχής στα οικονομικά θέματα, στον οικονομικό πλούτο. Είναι μια πλούσια χώρα το Ιράκ. Και όσον αφορά τον φυσικό πλούτο, τα ορυκτά, τα μέταλλα, ε, την, ε, τους νέους που έχουν ή το δυναμικό, όμως αυτό δεν κατανέμεται με τον πιο δίκαιο και ισοδίκαιο τρόπο. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να μπορέσουν με βάση την ένομη τάξη να λειτουργήσουν όλα αυτά, με, βάση, με βάση το Σύνταγμα. Και φυσικά σημαντικό άλλο αίτημα προ όλου, Αυτό αφορά την κυβέρνηση αλλά αφορά επίσης και την πλευρά των Σουνιτών. Η τάση ποια είναι να υπονομευθεί το κοινοβούλιο, να υπονομεύεται το κοινοβούλιο και να ε, απόσχουν από το κοινοβουλευτικό πλαίσιο, να υπονομεύουν το, τον Πρωθυπουργό και το, την κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδυναμώνει τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα, δεν τα ενδυναμώνει. Όταν λένε κάποιοι ότι ο ένα ή άλλο έχει πρόβλημα με τον Πρωθυπουργό. Συγγνώμη, ποια, ποια σχέση έχει αυτό με την ε, καμπάσα. Μπορείτε να μα πείτε, θα, θα έρθω σε αυτό το θέμα. Θα, θα έρθω σε αυτό αμέσω στη συνέχεια. Θα έρθω στο, στο θέμα καμπάσα σε ένα λεπτό. Η κύρια ανησυχία είναι ότι η χώρα αυτή βρίσκεται σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι, επικίνδυνο σταυροδρόμι και υπάρχει ο κίνδυνο να οπισθοχωρήσει σε μια έκρηθμη βία. Έρχομαι στην Καμπάσα τώρα και θέλω εδώ να ζητήσω την αρρωγή σας, τη βοήθειά σας στο Ιράκ να ενταχθεί σε ένα περιφερειακό πλαίσιο και να επανέλθει στην περιφερειακή αυτή συνιστόσα από πλευρά της διεθνούς κοινότητας. Αυτό θα ήταν το μήνυμά μου προς εμάς στο Ευρωκοινοβούλιο. Είδα πολλούς από εσάς χθε, αλλά επίσης και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Ε, στις 22 Απριλίου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εκφράζουν την ανησυχία τους, εκφράζουν την ανησυχία τους για την επιδείνωση της κατάστασης στο Ιράκ. Τώρα, το επόμενο πρόβλημα που έχουμε είναι το ζήτημα των σειράξεων Κούρδων Αράβων, που δεν έχει επιληθεί και αυτό λιμνάζουν τα πράγματα όσον αφορά τα εσωτερικά επίμαχα σύνορα. σύνορα. Δεν υπάρχουν συμπεφωνημένα σύνορα μεταξύ των περιοχών των Αράβων και της περιοχής των Κούρδων. Εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Εσωτερικά η κατάσταση καθορίζεται από την σύραξη Σουνιτών κατά της Βαγδάτης. Αλλά αυτό είναι επίσης και ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να θυμόμαστε. Έρχομαι στο θέμα Καμπάς, αλλά η ε, ενθαρρυντική παρατήρηση είναι ότι θα πρέπει οι σχέσεις του Ιράκ με το Κουβέιτ να μπορέσουν να εξομαλυνθούν. Είναι το κεφάλαιο 7. Να μπορέσει να ξεφύγει από τα ψηφίσματα του 7 η χώρα αυτή που θεωρείται επιβάρυνση στη χώρα, της χώρας αυτής από την περίοδο του πολέμου κατά του Σαντάμ Χουσέιν. Υπήρξε μια διμερή συμφωνία για τα σύνορα μεταξύ Ιράκ και Κουβέιτ. Υπάρχουν θετικές προοπτικές να βελτιωθούν οι σχέσεις, να βελτιωθεί η κατάσταση του Ιράκ σε σχέση με τις σχέσεις του, σχέσεις του Ιράκ προς το Κουβέιτ. Σύντομα να πω δύο λόγια τώρα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω το ανέφερα και την τελευταία φορά που είχα προσέλθει ενώπιόν σας. Εμείς από τα Ηνωμένα Έθνη είμαστε σχετικά μόνοι και απομονωμένοι στο Ιράκ. Χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα ένα σύμμαχο. Αυτός μπορεί να είναι μόνο ένα σημαντικός ισχυρός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αντιπροσωπείας σας, του πρέσβη σας στο Ιράκ, ώστε να, πάρουμε, να έχουμε πολιτική πολιτική παρουσία εκεί, ευδιάκριτη πολιτική παρουσία. Η πολιτική συμμετοχή είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντικό να ε, επικεντρωνόμαστε σε αυτήν. Όμως όλο και περισσότερο πιστεύω ότι είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρώνεται σε ένα πολιτικό ρόλο που θα ασκεί στο Ιράκ από κοινού μαζί μας των Ηνωμένων Εθνών, τους εκπροσώπους, διότι η καιροί είναι όλο και πιο κρίσιμη και όλο και πιο επικίνδυνη. Να μην απομονωθεί λοιπόν το Ιράκ από τις άλλες περιοχές και περιφέρειες ε, συζητάμε τη Συρία, το θέμα της Συρίας, αλλά όχι το Ιράκ. Είναι όμως δύο όψεις του ιδίου με, ε, νομίσματος να δούμε το σύνολο της περιφέρειας της περιοχής αυτής συνολικά, ολοκληρωμένα, να μην απομονωμένουμε τις δύο χώρες. Είναι δύσκολο βέβαια αυτό, είναι δύσκολο και για τα Ηνωμένα Έθνη. Όμως θα πρέπει μια περιφερειακή προσέγγιση να υιοθετηθεί για το Ιράκ, για το Λίβανο, για το Ιράν ώστε να μπορέσουμε να απαμβλύνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις των όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και τεκταίνονται σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Και καταλήγω τώρα στην ε, καμπάσα, διότι ξέρω ότι αυτό έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη πολλών από εμάς και σας απασχολεί ιδιαίτερα. Αυτό αυτή τη στιγμή ως θέμα βρίσκεται, ε, έχει ε, και αυτό παγώσει, έχει λιμνάσει και αυτό βρίσκονται στο Camp Liberty, Liberty ε, Πάμπολοι οι οποίοι ε, μεταφέρθηκαν εκεί και εξακολουθούν να βρίσκονται 100 περίπου στην Καμπάσα. Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δυσχερής, πιο δύσκολη με τους ε, Μουτζαχεντίν Χαλκί τους επαναστάτες του λαού. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα θέματα ε, MK e που έχουν δυσκολία να έρθουν σε επαφή και να συνεννοηθούν με τους Γιουνάμι. Επίσης όμως και δυσκολίες με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Ε, εν τω μεταξύ έχουμε τρεις ε, περιοχές μεταγκατάστασης ε, ε, προς την Αλβανία, 100 θα πάνε στην ε, Γερμανία. Η Ήπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και στο Camp Liberty με τις συνεντεύξεις για την επίλυση προβλημάτων, solutions interviews, πολλές φορές δεν εμφανίζονται πολύ. 34 ζητήθηκαν να προσέλθουν σε αυτές τις συνεντεύξεις, δεν πήγε κανείς. Έλλειψη λοιπόν συνεργασίας μαζί μας, έλλειψη συνεργασίας με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών, με τις αρχές διαχείρισης ε, διοίκησης του στρατοπέδου και όλο και μεγαλύτερα προβλήματα με τους επόπτες, monitors. Ξέρετε ότι χρηματοδοτεί 12 εκατομμύρια, με 12 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτή τη δράση συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ πάνω από 100 στελέχη UNAMI και άλλες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών εργάζονται σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της ΕΠΑ αυτή η πρωτοβουλία. Και είναι φυσική συνέπεια ότι στην ε, διεργασία μετεγκατάστασης που πρέπει να συνεχιστεί προς άλλες χώρες, έλλειψη συνεργασίας είναι η πρώτη μου λοιπόν παρατήρηση. Δεύτερη, η ε, εκένωση της Καμπάσα που ε, προαναγγέλθηκε από την κυβέρνηση. Όπως είπα, 100 βρίσκονται ακόμα ε, άτομα στην Καμπάσα. 100 έχουν ακόμα εκεί την έδρα τους. Επειδή πρέπει πρέπει να ε, διαφυλαχτεί, να διαφυλαχτούν ε, ε, περιουσιακά στοιχεία. Προσπαθήσαμε πολύ σκληρά από πέρυσι να ενθαρρύνουμε την ηγεσία του MK να διορίσει τρεις Ιρακινούς δικηγόρους για να επιληθούν τα προβλήματα περιουσιών. Αυτό ε, διαρκώς συνεχιζόταν και ε, από άλλες χώρες προσερχόντουσαν δικηγόροι στο Ιράκ. Ε, η ΕΜΚ e είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, θεωρεί η κυβέρνηση του Ιράκ. Και κάθε ελευθερία και κάθε έναν από αυτούς που βρίσκονται στο Ασάφα τους θεωρούν παράνομα εγκατεστημένους στο Ιράκ. Ο στόχος είναι λοιπόν να εκενωθεί αυτά τα άτομα από την Καμπάσα, εμείς προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση, όχι μόνο τους ενθαρρύνουμε, αλλά το λέμε και ξεκάθαρα να αποφευθεί οποιαδήποτε βία η λύση διότι αυτό θα καθιστούσε οποιαδήποτε επίλυση του προβλήματος ακόμα και δυσχερέστερη. Όμως θα υπάρξει δικαστική εντολή κατά το άμεσο μέλλον να εκτοπιστούν, να εκενωθούν οι υπόλοιποι 100 και να διοριστεί μια επιτροπή ώστε να αξιολογήσει τα θέματα περιουσιών, να καταγραφεί ένα μητρό να συνταθεί αυτών των περιουσιακών στοιχείων και είναι και το θέμα και των δικηγόρων που θα πρέπει να αποσταλούν και προς αυτή την Επιτροπή. Εμείς προσπαθούμε προσπαθούμε να αποθαρρύνουμε την κυβέρνηση του Ιράκ να μην αναλάβει οποιαδήποτε βίαιη δράση κατά του στρατοπέδου Ασάφ. Αλλά λέει η κυβέρνηση και δεν είναι η δική μας άποψη, η δική μου άποψη λέει η κυβέρνηση ότι μια και θεωρούν ότι βρίσκονται παράνομα αυτοί οι αλλοδαποί στη χώρα, τι κάνουν οι Ευρωπαίοι δεδομένη μια τέτοια κατάσταση. Δεν έχουμε εμεί το δικαίωμα να του εκτοπίσουμε, να του διώξουμε. Εμεί δεν παίρνουμε μέρο υπέρ καμιά πλευρά. Είναι ανθρωπιστικό θέμα. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε ούτε σε θέματα ιδιοκτησιών, ούτε σε άλλα θέματα. Θέλουμε το ανθρωπιστικό αυτό πρόβλημα να επιληθεί με ειρηνικό τρόπο. Και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι όλο και περισσότερο δύσκολο για μα να το αντιμετωπίσουμε το σύστημα εντολών και διακυβέρνησης στο ίδιο το στρατόπεδο Camp Liberty. Όλο και δυσχερέστερη η κατάσταση για όσους βρίσκονται εκεί. Υπάρχουν ε, διάφοροι τομείς, ε, έλλειψη ελευθερίας ε, κινήσεων, έχουμε εκθέσεις παρακολούθησης και εποπτείας πάνω από 300 από την έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας. Έχουμε πραγματικά μια επισκόπηση. Πώς λειτουργούν τα πράγματα σε σχέση με τη δομή εντολών και ε, διακυβέρνηση στο Camp Liberty είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα να ανεχθούμε πλέον ως καθεστώς. Απουσία ελευθερίας κινήσεων βρίσκονται σε κάποιους τομείς και δεν μπορούν ε, να συνέρχονται ελεύθερα και υπάρχει ένα αυστηρότατο σύστημα εποπτείας. Μετά το όριο, ε, οι περιορισμοί σε πρόσβαση, σε περίθαλψη υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικών υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στις κλινικές και σε ε, ιατρικό προσωπικό. Δεν πρέπει να παρακολύονται. Υπάρχουν πολλοί που είναι πάρα πολύ άρρωστοι, άλλοι που είναι παραπληγικοί και πλήττονται ιδιαίτερα από αυτή την κατάσταση και αξίζει να μπορούν να πηγαίνουν σε ένα νοσοκομείο ή να έχουν ιατρική περίθαλψη εφόσον το αξίζουν να το κάνουν και πρέπει να μπορούν να το κάνουν αυτό. Επόμενο θέμα, δεν υπάρχει ελευθερία επικοινωνίας, δεν υπάρχουν ελεύθερα τηλέφωνα για την επικοινωνία αυτών των ατόμων εκεί. Δεν υπάρχει ελεύθερο διαδίκτυο, δεν υπάρχει ελεύθερη τηλεόραση ή τηλεοπτικές εκπομπές και αυτό είναι κάτι που τον 21ο αιώνα είναι δεδομένο παντού. Ε, ε, δεν έχει πρόβλημα με το ελεύθερο διαδίκτυο η κυβέρνηση του Ιράκ, όμως κάθε ένας από όλους αυτούς θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα ελευθερίας να μπορούν να πηγαίνουν να ε, πληροφορούνται ελεύθερα χωρίς να παρακολύονται από τους επόπτες. Έχουμε όλο και δυσχερέστερες επαφές με αυτούς που βρίσκονται εκεί εμείς και αυτό είναι ένα θέμα των ε, ε, διαβουλεύσεών μας φυσικά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επόπτες μας ε, θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση και ελεύθερες συζητήσεις και συνεντεύξεις με τα άτομα εκεί. Αυτό είναι όλο και πιο δύσκολο. Είναι κάτι που παρακολύεται από τις δομές εποπτείας και ήδη είχαμε γεγονότα εχθές κιόλας όπου οι επόπτες διέκοψαν μια συνεδρίαση και δήλωσαν ότι ολοκληρώθηκε, λέει τερματίστηκε. Γιατί επειδή κάτι ήθελε να πει ένας από τους εγκατεστημένους εκεί που δεν ήταν της αρεσκίας τους και δεν έπρεπε να γίνει αυτή η παρέμβαση. Όλα αυτά τα γεγονότα καθιστούν ακόμα και πιο δύσκολο για όλους να έχουμε πρόσβαση σε αυτούς ε, τους ε, κατοίκους του Camp Liberty. Πρέπει να έχουμε ελευθερία πρόσβασης ε, και ελευθερία συνεντεύξεων και αυτό δεν διασφαλίζεται. Και αυτό είναι το ελάχιστο από πλευράς ανθρωπιστικού επίπεδου και ανθρωπιστικής βοήθειας. Όλοι να έχουν πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση και όλοι να μπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα αν θα μπορούν να φύγουν από αυτό το στρατόπεδο ή όχι. Ελευθερία κινήσεων. Συμπέρασμα τελικά. Πολύ συχνά γίνεται λόγος για το ότι θέλουν να επιστρέψουν στο Καμπάσαφ ε, οι ε, κάτοικοι αυτού, αυτού του Camp Liberty. Έχω έρθει σε επαφή και με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, μας λένε όχι, αυτή είναι η τελική διαχωριστική γραμμή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως πραγματικό πρόβλημα στο, του πραγματικού κόσμου. Δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουν στο Camp Ashafa. Δεν το επιτρέπει η κυβέρνηση. Να φύγουν από το Camp Liberty είναι η μόνη δυνατότητα να πάνε σε άλλες χώρες, σε τρίτες χώρες. Στην Αλβανία, Γερμανία. Σας ενθαρρύνω να έρθετε σε επαφή με την κυβέρνηση. Να στραφείτε στις κυβερνήσεις ε, ώστε να μπορέσουν ε, να γίνουν δεκτά αυτά τα άτομα στις χώρες σας ε, με μια μετεγκατάσταση. Η μετεγκατάσταση είναι η μόνη δυνατότητα δυνατότητα για να ε, μπορέσουν να διαφύγουν από αυτό το στρατόπεδο οι όσοι βρίσκονται εκεί. Ε, απευθύνω έκκληση να υπάρχει δυνατότητα να υπάρξουν αυτέ οι συνεντεύξει με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών. Όπω σα είπα, χθε δεν προσήλθε κανεί σε αυτή τη συνέντευξη έχουν φύγει 14 μέχρι την Αλβανία. Για την Αλβανία δεν επαρκούν με κανένα τρόπο αυτοί. Πρέπει να υπάρξει μια διοργανωμένη, οργανωμένη έξοδος αυτών των ατόμων προς τρίτες χώρες και στις 9 Φεβρουαρίου είχαμε ένα σημαντικότατο πλήγμα. Οκτώ που βρισκόντουσαν στο ε, στρατόπεδο αυτό δολοφονήθηκαν. Υπάρχει εδώ ευθύνη της κυβέρνησης του Ιράκ ε, για όσους είναι εγκατεστημένοι στο ε, στρατόπεδο Liberty. Δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει αυτές οι δολοφονίες. Διαμαρτυρηθήκαμε κάθετα και έντονα. Υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα προστατευτικά μέτρα τα οποία ζητούν να ληφθούν οι κάτοικοι, οι εγκατεστημένοι στο Camp Liberty. Αυτό το οποίο συνέβη το Φεβρουάριο δεν πρέπει πρέπει να με κανένα τρόπο ποτέ ξανά. Το τελευταίο πρόβλημα, αν επιτρέπετε το αναφέρω, είναι τα όσα γίνονται και λέγονται για τους εγκατεστημένους στο Liberty ή και στο Ashraf. Η επιστροφή στο Ashraf επεξήγησα ήδη. Απορρίπτεται από την κυβέρνηση του Ιράκ κάθετα. Δεν το δέχονται. Το άλλο είναι να ξεχωρίσουν οι Ιουνάμοι από το UNHCR, δηλαδή σε σχέση με την ύπατη αρμοστή από των Ηνωμένων Εθνών. Δεν γίνεται αυτό. το ε, μνημόνιο συνεννόησης ε, είχε υπογραφεί από κοινού. Δεν είναι δυνατό να υπάρξει ξεχωριστά ε, διαχείριση του χαρτοφυλακίου χωριστά του ενός από το άλλο. Πρέπει και τα δύο να εξεταστούν από κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δυνατότητα να παρέμβω πρόεδρε και ευχαριστώ για την προσοχή όλων σας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πρώτος που θα λάβει τον λόγο ο κύριος Στίβενσον, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Ιράκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αρχή της παρουσίασης του κύριου Κόμπλερ όταν έκανε μία αξιολόγηση της επιδεινούμενης κατάστασης στο Ιράκ. Είναι 700 θάνατοι οι οποίοι έλαβαν χώρα τον προηγούμενο μήνα και μόνον η συνεχιζόμενη ε, σύγκρουση ανάμεσα στις διάφορες ε, φατρίες ε, οδηγούμεθα σε έναν εμφύλιο πόλεμο εκτός και αν αναλυφθεί μια άμεση δράση έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση που να εκπροσωπεί όλο το λαό. Πάντως ε, θεωρώ ότι είναι κρίμα να κατηγορούμε και να είπε η κυρία Νάβη Πύλη στην Γενέβη για τις ε, εκτελέσεις ότι ήταν σαν να οδηγούνται ζώα προσφαγή. Εσείς στην ε, Βαγδάτη όμως κύριε Κόμπλερ δεν το είπατε αυτό. Εσείς είπατε ότι πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι ώστε να ε, εκπροσωπείτε και τα δύο μέρη και, τους, ε, και αυτούς που διαμαρτύρονται και βρίσκονται στο δρόμο κάθε Παρασκευή ε, και διαμαρτύρονται για την ε, βία της κυβέρνησης, αλλά ε, είπατε όμως ότι από πολιτικής πλευράς δεν μπορείτε να υιοθετήσετε τις θέσεις τους, γιατί πρέπει να εργαστείτε και με τις δύο πλευρές και με την κυβέρνηση. Όμως εγώ είδα ότι πολλοί από αυτούς ε, τους διαμαρτυρόμενους, ε, τους διαδηλωτές, ε, διαμαρτύρονται για την δική σας στάση, γιατί θεωρούν ότι συνεργάζεστε με την κυβέρνηση σε ορισμένα θέματα. Θέλω όμως να στρέψω την προσοχή μου στο τελευταίο κομμάτι της παρέμβασής σας για τα δύο στρατόπεδα, στο Άσραφ και στο Λίμπερτι. Είπατε ότι Έχουμε 3.100 άτομα από το Άσραφ που πήγανε στο Λίμπερντι και είπατε ότι τους μετακινήσατε ηθελημένα και υπογράψατε ένα μνημόνιο συνεργασίας μονομερός με την κυβέρνηση του Ιράκ χωρίς να συμφωνήσουν οι όσοι βρισκόντουσαν στο στρατόπεδο Άσραφ. Όμως κύριε Κόμπλερ ήρθατε εδώ και εδώ στο Κοινοβούλιο και φέρετε ένα ντοσιέ με φωτογραφίες που δείχνετε εμένα και άλλους ε, και άλλα εξέχοντα μέλη του Κοινοβουλίου ε, που, είχαμε, που βρίσκονταν στο στρατόπεδο, ε, στο Άσραφ, όπου ακούγαμε διάφορες υποσχέσεις ε, και εγγυήσεις ότι το στρατόπεδο είναι απόλυτα ασφαλές και τα λοιπά. Ο Ταχάδρα Μπεβέρνα, ε, ένας από τους υψηλούς αξιωματούχους της υπηρεσίας σας, ε, παρετήθηκε και όταν βρισκόταν με υπόρκο, είχε ορκιστεί ενώπιον της Γερουσίας, δήλωσε ακριβώς τα, τα αντίθετα. Δεν μπορώ να καταλάβω, φέρατε φωτογραφίες για να ε, κοροϊδέψετε τα μέλη του Κοινοβουλίου, αυτή είναι η προσπάθειά σας. Επομένως, όταν λέτε ότι υπήρξε μια υπέθεση τον Φεβρουάριο που πέθαναν 7 άτομα, όταν εσείς είπατε ότι η ασφάλεια αυτών των ανθρώπων στο, στρατόπεδο Λίμπερτι ήταν εγγυημένη, τότε γιατί τέσσερι μήνες αργότερα δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για τα 3.100 ε, άτομα, γιατί λέτε ότι διαμαρτυρηθήκατε εσείς ο, στην κυβέρνηση, εσείς ο ίδιος ε, αφήσατε ακάλυπτους αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, είπατε ότι δεν υπάρχει συνεργασία με, το, με, το, με τους πολίτες Άσραφα. Έχω εδώ πέρα όμως πολλά με ένα κατάλογο ατόμων εδώ. Κοιτάξτε, έχουμε 10 άτομα ακόμα που ζητάνε το λόγο και πρέπει να τους δώσουμε την δυνατότητα να μιλήσουν και να απαντήσει και ο κύριος Κόμπλερ. Äh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Εργάζομαι στην Επιτροπή, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα που εσείς μας δείξατε για την κατάρρευση διάλυση του Ιράκ. Υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις βασανιστήριων ε, στις ε, φυλακές. Είναι λοιπόν ευρύτατο αυτό το φαινόμενο. Ταυτόχρονα έχουμε και την Ανεξάρτητη Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσον μπορεί να εργαστεί αυτή για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα. Είπατε επίσης ότι δεν μπορεί απομονωμένα να εξετάζεται η περίπτωση του Ιράκ. Έχουμε τόσους ε, πολλούς ε, πρόσφυγες από το Ιράκ προς τη Συρία και αντίστροφα πρόσφυγες από τη Συρία προς το Ιράκ. Πώς έχει η κατάσταση για τους πρόσφυγες εκεί στο Ιράκ. Και τελευταίο, συζητήσαμε διεξοδικά για το Camp Ashraf. Όταν είχατε έρθει την τελευταία εδώ φορά, μας παρακαλέσατε θερμά στις χώρες μας να κάνουμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας, να γίνουν δεκτά άτομα στις χώρες μας, γιατί δεν είναι ασφαλή εκεί, όπως έδειξαν οι επιθέσεις σε αυτό το στρατόπεδο. με τώρα πάρα πολύ που λέτε ότι δεν υπάρχει, λέει, συνεργασία. Ακόμα και η δική μου κυβέρνηση ήταν πρόθυμη να δεχθεί άτομα. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο να επιτευχθεί αυτό. Το μας λέτε, να μας λέτε τώρα δεν υπάρχει πρόθεση ή προθυμία για συνεργασία είναι τόσο ασίδωτη και αθαίρετη η ηγεσία ώστε να μην υποστηρίζει μια τέτοια πρωτοβουλία. Ερώτηση υποστηρίζει την αντιπροσωπεία επιτόπου η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ. Yes, uh, thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απλώς να πω καταρχάς ότι χαίρομαι που έχουμε αυτή την ευρύτερη συζήτηση για το Ιράκ. Υπάρχουν ε, δυσκολίες, ε, ο ρόλος ε, του ΟΗΕ και Υπάρχει μια έκκληση όλο να παίξει ένα μεγαλύτερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε πώς οι Υπουργοί Εξωτερικών στο Συμβούλιο δεν κατάφεραν να αποφασίσουν κάτι ουσιαστικό για την ε, Συρία και πραγματικά χαίρομαι ε, γιατί ε, ακούστηκε αυτή η έκκληση σήμερα. Αυτό το οποίο σημαίνει ότι ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ένα πιο σημαντικό ρόλο. Τέλος πάντων, σε σχέση με αυτά που είπατε, ε, ε, καταλαβαίνω ότι δεν είσαστε ικανοποιημένο από όλα όσα γίνονται, από το επίπεδο δέσμευσης και τα λοιπά. Να είστε ειλικρινείς μαζί μας. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν μπορώ να καταλάβω... Αυτά αυτά τα ε, EMO, δεν ξέρω πώς θέλετε να τα πείτε, ακούστηκαν διάφορα ε, καταστροφικά αν θέλετε και κακά για, αυτές, ε, για, για αυτές τις, ε, αυτούς τους οργανισμούς. Ε, για άτομα τα οποία υπερασπίζονται αυτούς τους οργανισμούς, Καλό θα είναι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να δολοφονούμε αν θέλετε προσωπικότητες, ε, δεν μπορούμε να κατηγορούμε χωρίς στοιχεία ε, κάποιους ανθρώπους. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να είναι προσεκτικοί. Επίσης ο περιφερειακός χαρακτήρας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, εμείς συζητάμε κυρίως ας πούμε τη Συρία, το Μαυροβούνιο, μετά συζητάμε κάτι άλλο. Ε, πιστεύω ότι τα θέματα της, των θρησκευτικών διαφορών και τα λοιπά, ε, των επιμέρους διαφορών χάνονται γιατί εξετάζουμε στο σύνολο την χώρα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ε, προσέγγιση την, ε, που θα έχει περιφερειακό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στη Συρία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα. Λοιπόν, ο πρόεδρος ε, Παρέλ δίνει τον ε, λόγο, που έχει αναλάβει την, ε, την προεδρία δίνει το λόγο στην κυρία Γκόμες. Κύριε Κόμπλετς, θα ήθελα να μας πείτε πώς καταλαβαίνετε εσείς ε, τις συνέπειες της σύγκρουσης στην Συρία στο Ιράκ. Υπάρχει άμεση συνέπεια στην, σε αυτή την ολοένα αυξανόμενη βία που εμφανίζεται στο Ιράκ και κατά πόσον τα μέλη της κυβέρνησης, οι εκπρόσωποι των πολιτών, των διαφόρων εθνικών ομάδων, πώς, μπορούν να, πώς καταλαβαίνουν τις συνέπειες αυτές. Επίσης θα ήθελα να είστε πιο συγκεκριμένος όταν ζητάτε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ένα πιο έντονο πολιτικό προφίλ. Εγώ τη γνωρίζω, ε, την, την κυρία Γιάννα Εβάσκοβα, ε, την εκτιμώ ιδιαίτερα, πιστεύω ότι έχει το σωστό προφίλ, για το σωστό πολιτικό προφίλ το οποίο αναφέρεται και όντως θα πρέπει όλα τα, ε, όλες οι πλευρές από, του, του Ιράκ να ε, προσπαθήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους. Διότι ακριβώς και η Ευρώπη έχει κάθε συμφέρον να είναι δημοκρατικό και ενιαίο ενωμένο το Ιράκ ποιοι είναι οι περιορισμοί. Όταν ήμουν εισηγήτρια στο παρελθόν για το Ιράκ ε, και ε, έχω την έκθεση του 2008, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ε, η αυτοκίνηση αυτόνομη, ε, το, να έχουμε αυτόνομο χώρο αν θέλετε εμεί εκεί, δικός μου, δικό μας είναι δύσκολο, διότι είναι θέματα ασφάλειας. Αυτό είναι όμως το μόνο πρόβλημα. Για, τώρα για το MAK. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μέσω ε, ημών Πρόεδρε να ζητήσουμε από την κυρία Άστον να έρθει εδώ, διότι έχουμε 12 εκατομμύρια ευρώ των Ευρωπαίων φορολογουμένων που ξοδεύονται ε, για τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες. Βέβαια αυτό έχει και πολιτικές ε, συνέπειες, ε, διότι με τον τρόπο αυτό τα, όσοι ήταν στο στρατόπεδο Ασράφ έπρεπε να μεταφερθούν σε ασφάλεια και υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν μπορούν να επιστρέψουν στο Ιράκ. Όμως η πολιτική εξουσία παρεμποδίζει την, το έργο αυτό, όπως μας είπε και ο πρέσβης κύριος Κόμπλερ και θέλω ακριβώς να ακούσω από την κυρία Άστον ποιος φταίει. Θέλω να αναλάβει τις ευθύνες. Γιατί και από τα Ηνωμένα Έθνη και από την αντιπροσωπεία των, των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θέλω να καταλάβω πώς ε, επιτρέψαμε να γίνει κάτι τέτοιο. Όσοι ήταν στο στρατόπεδο Ασραφ δεν είχαν την ευκαιρία, δεν είχαν το δικαίωμα να μιλήσουν ε, στους εκπροσώπους της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους, τους πρόσφυγες, χάρη. Ε, επίσης να σας πω ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά τα που είπαν πολλοί από τα μέλη της, ε, του, του Κοινοβουλίου. Δηλαδή το, όπως έκανε παραδείγματο χάρη η ε, πρόσωπος Επιτροπής ε, για το Ιράκ που κατηγόρησε, ε, σας κατηγόρησε και προσπαθεί να σας να υποβαθμίσει το, το έργο σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούκαν είναι ο επόμενος ομιλητής και ρωτώ επομένως. Ε, σε σχέση με αυτά που είπε και ο κύριος Στίβενσον, μία πάρα πολύ προσωπική παρέμβαση κύριε Πρέσβη, την οποία κατέγραψα όταν μιλούσατε για τις συνθήκες ε, διαβίωσης ε, στο στρατόπεδο Άσραφ και στο στρατόπεδο Λίμπερτι και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Συμφωνώ μαζί σας ε, όσον αφορά τις κακές συνθήκες διαβίωσης. Δεν έχουν ε, θέματα τα οποία ε, δεν έχουν υπηρεσίες τις οποίες εμείς θεωρούμε αυτονόητες. Όμως, μου ακουστήκατε σαν ένας αντικειμενικός παρατηρητής ενώ πιστεύω ότι είναι δική σας ευθύνη κύριε πρέσβη να προσπαθήσετε να βοηθήσετε να βοηθήσετε αυτούς που ζουν σε αυτά τα στρατόπεδα. Αυτή ήταν η παρατήρηση που θα θέλω να κάνω κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρέσβη, συγγνώμη. Ο κύριος Λαντσμπέργκης είναι ε, ο καλός μου γείτονας, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Κόμπλερ, υποστηρίζετε την έκκληση να γίνει ε, να γίνει μια έρευνα για τις ε, ενέργειες του πρέσβη Κόμπλερ και των ε, συνεργατών του για, την, για τα όσα έκαναν στο στρατόπεδο Άσραφ. Στις Ε, σε 27 Μαΐου πολλοί, ε, όπως ο πρόεδρος Ομπάμα, ο Γενικός Γραμματέας Μπάνκι Μούνα και άλλοι, είπαν ότι θα έπρεπε να γίνουν έρευνες. Και αυτή η έρευνα πιστεύω ότι θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει το όνομά σας από πολλές κατηγορίες ε, για κακοδιαχείριση. Επομένως ρωτώ, θα ζητήσετε να γίνει μια Έχετε ζητήσει ήδη μια τέτοια έρευνα ή απλώς περιμένετε υπομονετικά το τέλος της αποστολής σας για να εγκαταλείψετε το, την Βαγδάτη χωρίς ε, να λογοδοτήσετε. Και ε, η, η, το έργο σας ε, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και καταστροφικό, διότι δεν μπορέσατε να μεταφέρετε με ασφάλεια εξέχοντα ε, μέλη της ε, Ιρακινής ε, κοινωνίας. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα. Χρησιμοποιήθηκε ο εκπρόσωπος του Ηνωμένων Εθνών για να ικανοποιηθούν συμφέροντα ξένων χωρών ε, όσον αφορά την ε, μεταφορά των προσφύγων. Πρόεδρε, για την εδαφική ακαιρεότητα του Ιράκ. Είστε πολύ κοντά και έχουμε φτάσει πολύ κοντά στην διάλυση της χώρας. Δεν έχει ξεκινήσει όμως η διαδικασία ακόμη. Ανακοινώσατε την επιστροφή Κούρδων βουλευτών στην ε, Βαγδάτη. Όμως η στάση της κυβερνώσας πλειοψηφίας κατά των Σουνιτών είναι εκτός από κάθε λογικό πλαίσιο. Περιμένω λοιπόν κάποια ανακοίνωση, γιατί είπατε ότι θα θέλετε να δημιουργηθεί καλύτερο κλίμα για το μέλλον. Αλλά δυστυχώς το πολιτικό περιθώριο, το πολιτικό σκηνικό μάλλον είναι τόσο δηλητηριασμένο που θα πρέπει να αναζητήσουμε διαφορετικά και σε εναλλακτικέ και σενάρια. Έχω λοιπόν πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Θα πετύχουμε κάτι χειροπιαστό, το οποίο πραγματικά να ενδυναμώσει τι δημοκρατικέ δυνάμει. Θα ε, προσφέρουμε τα εργαλεία για να επικοινωνήσουμε με τον Πρωθυπουργό Μαλίκη. Θα τον διαβεβαιώσουμε ότι θα ε, αποτρέψουμε συμπεριφορές που έχουμε δει ως τώρα να λαμβάνουν χώρα. Τι θα γίνει με το διορισμό υπουργών του Υπουργού Εξωτερικών, ε, εσωτερικών μάλλον Υποθέσεων και Άμυνα, που δεν έχουν διοριστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να. Ο κύριο Τέρχο, μάλλον. Θέλω και εγώ να παραμείνω στα θέματα ασφάλεια. Μιλήσατε για την ε, βομβιστική επίθεση και τι τρομοκρατικέ επιθέσει γενικότερα. Μετά από τόσου μήνε όλες οι βελτιώσεις που θα μπορούσαν να έχουν επιφερθεί δεν έχουν ε, περατωθεί. Γιατί δεν βοηθάτε τους ανθρώπους στον καταβλισμό Liberty και με την αποκομιδή τομάτων. Και γιατί οι συνθήκες ασφαλείας δεν έχουν ε, βελτιωθεί αρκετά ακόμα. Παρακαλώ πείτε μας γιατί. Ευχαριστώ πολύ. Μια παρατήρηση. Η κανονική, ο κανονικός πληθυσμός του Ιράκ βρίσκεται υπό απειλή όπω κανένας άλλο πληθυσμό. 700 Ιρακινοί, όχι στο, στο Καμπάσα ή στο Καμπλίμπαρτι, τον Απρίλιο 700 Ιρακινοί σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να δούμε στη συνολική εικόνα. Ο κύριος Κόμπλερ έχει το καθήκον να δώσει τη συνολική εικόνα και όχι μόνο να περιορίζεται στο Καμπλίμπαρτι η κατάσταση στη συνολική αυτή χώρα, η συνολική κατάσταση είναι ολέθρια. Δεν είναι η ενοχή των Ηνωμένων Εθνών αυτή η κατάσταση. Άλλοι είναι ενόχη γι' αυτό. Εσείς έχετε τον λόγο τώρα παρακαλώ. Thank you, Mr. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά αν επιτρέπετε στην παρέμβασή μου. Λοιπόν, στα Ολλανδικά θα μιλήσω και θα ήθελα για άλλη μια φορά να επιστήσω την προσοχή στην κατάσταση στο Κουρδιστάν, στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Γνωρίζετε ότι έχουμε και τις ε, περιφερειακές εκλογές που έγιναν στις 20 Απριλίου. Είχαμε 18, 12 ε, ή 18 εκλογικές περιφέρειες. Αυτό που με ξέπληξε περισσότερο ήταν ότι είχαμε εκλογές και σε άλλες ε, περιοχές επίσης αυτή της ευρύτερης ε, περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν. Βλέπουμε ότι Ντεγιούρε είναι μέρος του Ιράκ αυτή η επαρχία, όμως ε, πρακτικά είναι ανεξάρτητη. Υπήρξαν διαφορετικές εκλογές που διεξήχθησαν εκεί και διαπιστώσαμε ότι αυτή η περιοχή de facto όλο και περισσότερο είναι ανεξάρτητη και γίνεται κάθε μέρα και περισσότερο ανεξάρτητη. Υπάρχει για παράδειγμα μια αγορά εξαγωγών ε, πετρελαίου του, που είναι προ προμηθευτεύων προϊόν του Ιρακινού Κουρδιστάν. Θα ήθελα να ξέρω το εμπόριο με την Τουρκία διασφαλίζει ή όχι την ενότητα της χώρας, την υπονομεύει μήπως. Και θα προσθέσω τη φωνή μου σε σχέση με την ασφάλεια των προσφύγων. Και έχω υπόψη εδώ φυσικά την κλιμάκωση της βίας σε σχέση με έναν εμφύλιο πόλεμο που είναι μια πιθανή προοπτική. Θέλω να ξέρω ποιε επιπτώσεις θα είχε κάτι τέτοιο. ποιε επιπτώσεις θα είχε στην ανθρωπιστική κατάσταση, για παράδειγμα των ε, σύρων προσφύγων. Ποιε επιπτώσεις θα υπάρχουν σε σχέση με αυτή την εμφύλια σύραξη της Συρίας στι όμορε χώρε στην Ιορδανία. Ποιε επιπτώσεις θα υπάρχουν, διότι είναι γειτονικέ χώρες αυτές και χώρες όπως η Ιορδανία δεν μπορούν περισσότερο να αντέξουν μια τέτοια κατάσταση και αυτές θα απορροφηθούν σε μια τέτοια σύραξη. Ευχαριστώ. Um- Σα ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για το ότι καθυστέρησα και δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω όλη τη συζήτηση, αλλά ένα μέρος της μόνο. Ίσως απαντήθηκε το ερώτημά μου, το ερώτημα το οποίο μόλις θα διατυπώσω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε πραγματικά στο ότι οι άνθρωποι στο ΚΑΠ και να μπορέσουν να βρουν άλλες χώρες, να πάρει σε ένα ασφαλές ε, περιβάλλον, σε ένα ασφαλή περίγυρο. Υπάρχουν προσπάθειες να εξευρεθούν χώρες υποδοχής. Ίσως απαντήσατε αυτό το ερώτημα. Πόσοι από αυτούς ενδυνάμει μπορούν να μετεγκατασταθούν αλλού Ποιε διασφαλίσει έχετε από άλλε χώρε, για πόσε χώρε κάνουμε λόγο για αυτή τη μετεγκατάσταση αυτών των ανθρώπων. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Να πάνε σε ασφαλεί χώρε, ευρωπαϊκέ χώρε ε, τα άτομα αυτά. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτό το οποίο συμβαίνει στο Ιράκ. Το πρόβλημα δεν είναι όμω οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτά τα στρατόπεδα, αλλά η ηγεσία των Ιρακινών που δεν έχει κανένα συμφέρον να πάνε καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με αυτού του ανθρώπου, γιατί θα χάσει τον έλεγχο επ' αν πάνε στην Ευρώπη και σε ασφαλεί χώρε. Θέλω να συνεχίσετε την προσπάθειά σα εξευρεθεί μια ασφαλής χώρα υποδοχής για αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είναι εύκολο να συνεχίσω, διότι θα ήθελα και εγώ να απευθύνω την ίδια έκκληση με τον προλαλήσαντα. Ε, ανησυχώ ιδιαίτερα για την κατάσταση στο Ιράκ και για την ε, πιθανότητα επιδίνωσης της κατάστασης αυτής. Κύριε Κόμπλερ, φαίνεται ότι είσαστε ένα αμφιλεγόμενο άτομο στο Ιράκ, διότι κάποιοι ε, Ιρακινοί ε, σας λατρεύουν, ε, άλλοι ζητάνε την παρέτησή σας, π.χ. ο αρχηγός ε, της αντιπολίτευσης, ο οποίος λέει ότι είσαστε πολύ κοντά στην, στις θέσεις της κυβέρνησης, εσείς λέτε ότι μπορείτε, προσπαθείτε να κρατήσετε μια κάποια απόσταση, όμως το πρόβλημα είναι, το ανθρωπιστικό πρόβλημα υπάρχει με το στρατόπεδο Liberty. Ας αφήσουμε τις, τους πολιτικούς λόγους, έχουμε πάνω από 3.000 άτομα εδώ και δεν μπορούμε και εσείς δεν μπορείτε να προσφέρετε κάποια λογική απάντηση όσον αφορά την ασφάλειά τους. Ε, εσείς ε, διαμεσολαβήσατε για την ε, μεταφορά τους, Είσαστε υπό το, είχαμε τον έλεγχο και την πίεση της Ιρακινής κυβέρνησης, αλλά εσείς είπατε ο ίδιος ότι η ασφάλεια τους ήταν διασφαλισμένη. Τώρα κανείς δεν μας αγγιάται ότι η επίθεση που έλαβε χώρα δεν θα ξαναλάβει πάλι χώρα και το 80% ή ε, της ευθύνης είναι ανήκει σε εσά. Επομένως, θα πρέπει να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας ε, έτσι ώστε να ε, διορθωθεί η κατάσταση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να βρούνε μια λύση. Όλοι μαζί πρέπει να τη βρούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και συμφωνώ ότι όπως αυτό το, το πρόβλημα με αυτήν την, ε, του είδους τη συνάντηση είναι ότι εμείς κάνουμε πολλές ερωτήσεις, λέμε, κάνουμε παρατηρήσεις και μετά όποιος, αναλάβει, όποιος είναι στην έδρα δεν θα αφήσει τον κύριο Κόμπλερ να απαντήσει. Λοιπόν, έγινε μία, ε, είπατε για ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων ο οποίος μεταφέρθηκε στην Αλβανία. Ε, δεν ήταν όσο είπατε. Τώρα, επίσης η κατάσταση επιδεινώνεται, δεν βελτιώνεται. Δικό, δική, σας, δική σας ευθύνη είναι. Για, το, για τα στρατόπεδα, το στρατόπεδο Άσραφ η κατάσταση είναι τραγική, πρέπει να γίνουν και έρευνες Είπατε ότι η κυβέρνηση θεωρούν, θεωρεί ότι τα 100 άτομα τα οποία βρίσκονται στο, στην Άστραφη είναι τρομοκράτες. Από εδώ έχουν αποχαρακτηριστεί από εμά. Από του Αμερικανού έχουν αποχαρακτηριστεί σαν από τρομοκράτε και δεν μπορείτε να πείσετε εσεί στην κυβέρνηση του Ιράκ ότι δεν είναι τρομοκράτε. Μα είπατε κάτι επίση ότι το δικαστήριο δεν μπορεί να τους ε, ε, να βγάλει μια απόφαση για να, τους, για να μετακινηθούν. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, διότι είχαμε τις επιθέσεις το Φεβρουαρίου, ε, η οποία μπορεί να επαναληφθεί και λέτε ότι δεν υπάρχουν και οι ιατρικές υπηρεσίες. Επίσης είπατε ότι δεν υπάρχουν κινητά τηλέφωνα. Λοιπόν, τι έχετε να μας πείτε, τι έχετε να δείξετε για το, έργο, για το έργο σας και κυρίως στο τέλος της ημέρας τα πράγματα είναι τραγικά θα έλεγα εγώ. Και ξέρω ότι αν είχα την πλειοψηφία στο Συμβούλιο Ασφαλείας που δεν την έχω τέλος πάντων θα σας είχα απολύσει. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Κόμπλερ, όπως ο κύριος Λάμσντορφ, ο συμπατριώτης σας, δεν είμαι υπέρ σας, αλλά κανείς δεν είναι τέλειος. Πριν από δύο χρόνια είχατε έρθει στο Ευρωκοινοβούλιο και με τις τότε εξελίξεις είχατε κάνει δύο βασικές υποσχέσεις. Ότι ο καταβλισμός Λίμπερτι θα είχε τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης όπως ο Ασράφ και ότι θα στέλνονται οι πρόσφυγες, αρκετοί από αυτούς, σε τρίτες χώρες που θα ήταν ασφαλέστερε και από τον καταπλημάσιο. Τώρα μα. Τότε μας είχατε δείξει υπέροχε φωτογραφίες του Μας είχατε παρουσιάσει μια υπέροχη εικόνα για το τι ωραίο μέρος θα γίνει το κατα... ο καταπλησμό Λίμπερτι. Τίποτα από αυτά δεν πραγματοποιήθηκε. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι κάτοικοι του Άσραφ δεν σας πιστεύουν. Δεν μπορείτε να είσαστε εμπλεκόμενος στην σύγκρουση και να είστε πιστικός προς τους πρόσφυγες. Είσαστε περισσότερο μέρος του προβλήματος παρά της λύσης. Δεν πιστεύετε ότι ήρθε η στιγμή να παρατηθείτε. I will be very brief. Ευχαριστώ, Έλμαρ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Κατά πρώτον, νομίζω ότι είναι πολύ κρίμα τέτοιες συζητήσεις να επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Κρίμα είναι αυτή η εξατομίκευση. Θα πρέπει να συζητάμε για τους 300.000 ανθρώπους που δεν μπορούν να ορίσουν τη μοίρα τους. και ακόμη και αν κάποτε ήταν ε, ένοπλοι πολεμιστές, τώρα δεν είναι. Αλλά μιας και είστε ο ειδικό εκπρόσωπος του ΙΕ, πρέπει να σας ρωτήσω το εξής. Τι θα κάνει ο ΙΕ για να λύσει έστω και το απλό βασικό πρόβλημα της ασφάλειας. Ο κύριος Ντέρμοντ είναι πρώην ειρηνευτής ε, διαπραγματευτεί για θέματα ειρήνευση. Δεν είναι δύσκολο να δώσετε στου ανθρώπου αυτού ε, κράνη. Και ο ΙΕ είναι υπεύθυνο εδώ, γιατί ήταν μέρο τη συμφωνία. Οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν αλλού. Δεν σα ρωτώ λοιπόν κάτι προσωπικό. Σα ρωτώ υπό την ιδιότητά σα ω προσώπου ενό διεθνού οργανισμού. Τι θα κάνετε για να αγγίθετε την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων. Κύριε Κόμπλερ, Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω με τις πολιτικές παρατηρήσεις πρώτα απ' όλα κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι εκτελέσεις. Ο κύριος Στίβενσον είπε γιατί δεν κάνατε τίποτα για να εμποδίσετε τις εκτελέσεις. Δεν το γνώριζα κύριε Στίβενσον. Το έμαθα τα ανακοινοθέντα στον τύπο. Το ξέρετε, είμαι βέβαιο ότι και εσεί το ξέρετε, ότι πριν, δύο μέρε πριν, από την υπόθεση ε, ε, ξε, καταδίκασα τι έξι αυτέ εκτελέσει και ζήτησα να υπάρξει και ε, μνημόνια κατανόηση για την κατάργηση τη ε, θανατική ποινή. Η, η υπόθεση Πιλάη προέκυψε αργότερα. 21 εκτελέσεις, συνοπτικές. Ναι, θανατώθηκε σαν ε, να ήταν ζώο σφαγείο. Έτσι έγινε. Αλλά Έκτοτε πόσες εκτελέσεις έλαβαν χώρα στο ε, Ιράκ. Μόνο εκείνες που ακολούθησαν αμέσως μετά και καμία άλλη. Κύριε Στίβενσον, ξέρετε ότι είναι καλύτερο να είναι κανείς διακριτικός. Ε, είναι καλύτερα να μην κάνει μεγαλόστομες δηλώσεις και να σώζει ανθρώπινες ζωές, παρά να κάνει το αντίθετο και να, βάζει, να κολλάει στον τοίχο την κυβέρνηση και να συνεχίζονται οι εκτελέσεις. 500 άτομα περίμεναν να θανατωθούν. Αλλά νομίζω ότι ήμασταν αρκετά ε, αποτελεσματικοί εγώ και οι συνάδελφοί μου, γιατί αυτή τη στιγμή, de facto, δεν υπάρχει καμία πολιτική υπέρ των εκτελέσεων στο Ιράκ. Αυτό μπορεί να πάψει αύριο, αλλά αυτό συμβαίνει και αυτό είναι μέρο τη δική μα εντολή και επιτυχία. Δεύτερο στοιχείο, βασανιστήρια. Κύριε Λόχμπιλερ, τα βασανιστήρια για κατάσταση στι φυλακέ. Το ίδιο ισχύει. Έχουμε σαφέστατη, ρητή και ηχηρή πολιτική υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μέρος των προτεραιοτήτων μας. Το λέω εδώ και το λέω στο, κάθε τηλεοπτική κάμερα και κατά πρόσωπο στους πρωθυπουργούς που συνάντησα και το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μία υπόθεση και μόνο βασανιστήριων είναι πάρα πολύ η κατάσταση στις φυλακές είναι φρικτές, είναι φρικτή. Βεβαίως ε, τα πράγματα αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Βεβαίως μιλώ κατά της παραβιάσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι είμαστε μου Μουτζαχεντίν. Οι άνθρωποι στις φυλακές, οι ε, βίες αποσπάσεις ομολογιών, τα βασανιστήρια, όλα αυτά είναι πράγματα που καταδικάζονται διαρκώς από μένα και από τους συναδέλφους μου και το κάνω διαρκώς και κατά πρόσωπο με τους ισχυρούς όταν βρίσκομαι στην παρουσία του. Δεν είναι αυτά τα θέματα τα οποία ήρθαμε εδώ να λύσουμε. Δεν είμαστε σιωπηλοί. Κάθε περίπτωση ε, βασανισμού είναι η ε, περίπτωση που δεν έπρεπε να υπάρχει. Αλλά στη βελτίωση των συνθήκων τη φυλακή. Τι να κάνουμε, πώ στην πράξη να σταματήσουμε τα, βασανιστήρια, πώ να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώ θα μειώσουμε τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι μόνο θέμα βούληση, είναι και θέμα πράξεων, ενεργειών, δράση. Οι πρόσφυγες, εντάξει, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μιλήσατε για τους 3.200 έχουμε 1,3 εκατομμύρια εκτοπισμένους εσωτερικώς στο Ιράκ, 150.000 Σύρους προσφύγους και τίθεται θέμα ασφάλειας για τους 100.000 πρόσφυγες που έρχονται από τη Συρία. Είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα και αυτή για μας. Βεβαίως υπάρχουν καταβλισμοί κοντά στα σύνορα, τα οποία μπορεί να πληγούν από τους βομβαρδισμούς εδώ στην, και από τα πειρά ε, στον τομέα των προσφύγων και στην ανθρωπιστική μας ατζέντα, προφανώς αυτό είναι πρώτο σημείο και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Το θέμα της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε θα ήθελα να απαντήσω πολύ ξεκάθαρα εδώ. Εκτιμώ ιδιαίτερος τη δουλειά της πρέσβεως της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ ικανή, είναι πρώην συναδελφός σας και βλέπετε τι προσέγγιση έχει ακολουθήσει. Όμως το θέμα είναι τι περιθώριο υπάρχει. Και εκείνη το ξέρει και εμείς το καταλαβαίνουμε. Τι περιθώριο υπάρχει σε σχέση με την κυβέρνηση και τους υπολείπους, ώστε να μπορέσει να αναλάβει δράση και να έχει πολιτική ε, βαρύτητα. Εδώ έχουμε στενές επαφές και είναι πολύ σημαντικό εκείνη να πάρει τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τους πάει στους πρωθυπουργούς, στους ε, υφυπουργούς, ε, στους προέδρους του Κοινοβουλίου και το έκανε. Τέσσερι-πέντε μήνε πριν ξεκίνησε, ε, άρχισε να συμμετέχει ενεργώ και να επικοινωνεί, να περνάει τα μηνύματά μα. Όχι μόνο την, το διάβημα για την θανατική ποινή που ήταν πολύ ισχυρό, αλλά να περνάνε και πολιτικά μηνύματα μαζί με το κύρος των πρέσβειων της Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους παίρνει μαζί, τους, μαζί της και λέει, «Ε, πρόεδρε ε, του κοινοβου, της Βουλής, πρωθυπουργέ, έχετε ευθύνη εσείς ως πολιτικοί άνδρες για να μην καταρρεύσει η χώρα. Αυτό θα πει προβολή. Και αυτό θα πει επικοινωνία Προ την κοινή γνώμη. Τώρα, για τους υπόλοιπου τομεί. Ε, τον αναπτυξιακό, σημειώνω την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σταδιακή αποχώρηση, αλλά θα έπρεπε να είμαστε επιτυχεί εδώ και να υπάρξει ένα διάδοχο πρόγραμμα Επιτυχέ μάλιστα. Θα ήθελα να είμαστε πολύ πιο δραστήριοι στην εξέβρεση προγραμμάτων εδώ. Τι θα γίνει με, τις με το δικαστικό σύστημα, με τα σαφρονιστικά ιδρύματα, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ μπορούν να κάνουν κάτι εδώ. Την εκπαίδευση των ε, κρατουμένων, μάλλον όχι των ε, κρατουμένων, των ε, υπευθύνων των σοφρονιστικών ιδρυμάτων. Βελτίωση συνθηκών διαβίωση στι φυλακέ. Αυτά είναι πράγματα που εμεί μπορούμε να τα κάνουμε μόνο. Τέσσερι-πέντε φυλακέ πρότυπα θα ήταν ήδη μια αρχή. Η προβολή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εικόνα της και το κοινοβούλιο στο Ιράκ δεν έχει αυτή τη στιγμή καμία αξία. Μποϊκοτάρονται πολλά πράγματα λόγω της διαφορετικής μας ατζέντα, πολλά πράγματα δεν υλοποιούνται και ε, οι Ιρακινοί αυτή τη στιγμή έχουν τον περιδιευθύνη του στην πολιτική τελμάτωση. Οι διακοινοβουλευτικέ σχέσει τώρα, εσύ ίσω βουλευτέ, νομίζω, καλό θα ήταν, θα ήταν καλή ιδέα να ε, ξεκινήσετε και να αρχίσετε να συνομιλείτε με του ομόλογου βουλευτέ σα στο Ιράκ. Εσεί, ε, διακοινοβουλευτικό, θα μπορούσατε να καθορίσετε ένα πρόγραμμα δράση. Να όμω που είναι η δυσκολία όποτε μιλώ για το θέμα αυτό μου λένε ναι, αλλά η μόνη η, το μόνο σημείο στην ε, ατζέντα είναι ο Ασάφ. Καταλαβαίνω εδώ τη συγχύσή σα, καταλαβαίνω την ε, ε, ματέωσή σα λόγω τη έλλειψη πρόοδου. Το καταγράφω, αλλά δεν είναι το μόνο σημαντικό αυτό. Σε σχέση με το Ιράκ, έχει μονοπολίσει την προσοχή και έχει κρατήσει σε ομοιρία τη σχέση σα με την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο τη χώρα. Και αυτά λαμβάνουν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία, διότι έχουν δημοκρατική λειτουργία. Για να ξεφύγουμε λοιπόν από αυτήν την μονομερία προσέγγιση ε, για το Ιράκ, επικεντρωθήκε και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διαφθορά και στα βασανιστήρια και σε όλα αυτά τα θέματα μαζί με τους βουλευτές του Ιράκ και όχι μόνο με τον ε, Ασάφ, ο οποίος έχει παραμερίσει όλα τα άλλα σημαντικά ζητήματα για το θέμα του Κουρδιστάν και την Τουρκία. Αν θέλετε τη δική μου ειλικρινή εκτίμηση, δεν πρόκειται να καταρρεύσει το κράτος, ούτε θα υπάρξει δήλωση αναξαρτησίας στο εγγύς Η χώρα, το Κουρδιστάν, θα μείνει εντός του Ιράκ. Οι βουλευτές, οι Κούρδοι βουλευτές, τα μέλη της κυβέρνησης ξαναγύρισαν στη Βουλή προκειμένου να συμβάλλουν στις πολιτικές ε, συζητήσεις. Οι σχέσεις με την Τουρκία είναι πολύ καλές. Οι σχέσεις ε, του πρόεδρου Μπαρζάνη με την Τουρκία είναι καλές. Υπάρχει φυσικά και το θέμα του ΠΚΚ. Με το ΠΚΚ να επιστρέφει από το Μάιο, αυτό είναι καλό δείγμα και η ακεχηρία ε, φέρνει ειρήνευση, φέρνει ηρεμία στις σχέσεις μεταξύ Κούρδων της, Βα... Βαγδάτης και των Τούρκων. Η σχέση των Κούρδων με τη Βαγδάτη όμως, αυτές αυτές είναι το πρόβλημα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιωθεί. Και εδώ χρειάζεται η δική σας βοήθεια, διότι εσείς έχετε επαφή με τους βουλευτές του Κουρδιστάν. Με αυτούς πρέπει επίσης να συνομιλήσετε, διότι αυτή τη στιγμή σκοπεύουν να αναβάλουν τις εκλογές. Δεν μπορούν να αναβάλουν τις εκλογές τώρα μόνο και μόνο γιατί είναι ακόμα αισθάνεται ότι είναι αδύναμο και θα ανεβάλει για ένα εξάμεινο τις εκλογέ. Όχι. Είμαστε πολύ αδύναμοι όμω ακόμα. Πρέπει να ασκήσουμε το νόμιμο κύρος μας και να πιέσουμε τους βουλευτές. Πρέπει να τους πιέσουμε να γίνουν οι εκλογές. Πρέπει να ασκηθεί πολιτική πίεση και να μην υποκύπτουν σε άλλες πολιτικές ανάγκες. Χρειαζόμαστε εδώ τη στηρίξη και τη βοήθειά σας. Ο αντίκτυπος στη Συρία. Ή ο αντίκτυπο τη Συρία στο Ιράκ. Ε, πρέπει να πω ότι πολλά από τα προβλήματα στο Ιράκ προέρχονται από το εσωτερικό της χώρας. Εκείνοι τα προκάλεσαν. Εάν ήταν ήρεμη η Συρία και το Ιράν, δεν θα ήταν όλα ήρεμα. Τα εσωτερικά σύνορα δεν υπάρχουν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν προστατεύονται. Η διαφθορά θα σοβούσε. Οι οικονομικές πολιτικές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έκρηξη τον ε, τομέα της δημόσιας αυτά είναι άσχετα από τη Συρία. Η Συρία προφανώς και πυροδοτεί και ε, υποδαβλίζει όλα αυτά τα προβλήματα και επηρεάζεται το Ιράκ από τις εξελίξεις στη Συρία. Το θέμα είναι εάν μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή ώστε να έρθουν οι δύο πλευρέ μαζί και να συνομιλήσουν. Για την περιεφηροποίηση των Σουνιτών αυτό είναι σημαντικότατο, διότι το αίτημα μα προ την κυβέρνηση είναι να λάβει τα αιτήματα πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν μεροληπτούμε εμεί, είτε είναι θεμητά είτε όχι με την. Ε, ε, εξαίρεση τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί λαμβάνουμε θέση ε, και έχουμε πολύ σοβαρέ απόψει. Αλλά το ζητούμε να λάβουν σοβαρά υπόψη τα αιτήματα. Κανείς δεν έχει όφελος, όλοι τρομοκρατούνται από την προοπτική να επανέλθουμε σε καταστάσεις εμφύλιου πολέμου. Όπως τα προηγούμενα χρόνια 2006-2007. Εντάχει, για τον καταπλησμό Άσαφ, ξέρετε όλοι το ιστορικό. Το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει διότι υπήρξε πιεστική ανάγκη. Ο στρατός ήθελε να πάει στον καταπλησμό Ασράφ, όπου 3.200 άνθρωποι κατοικούσαν από το Δεκέμβριο του 2011 και ήταν υπουργική απόφαση της κυβέρνηση να κατακτηθεί αυτός ο καταβλισμό με τη βία. Αυτό είχε, απόπειρα, είχε γίνει απόπειρα για κάτι τέτοιο άλλες δύο φορές στο παρελθόν. 45 άνθρωποι πέθαναν για αυτό το λόγο το 2009 και το 2011. Τα ξέρετε, τα ξέρετε. 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ποια κατάσταση λοιπόν ε, διαμορφώθηκε. Προσπαθούμε να βρούμε διέξοδο. Δεν παίρνουμε εδώ πολιτική, δεν τοποθετούμαστε πολιτικά είναι τρομοκράτε ή όχι. Όχι, είναι άνθρωποι. Πάνω από όλα είναι άνθρωποι και αυτή η αποστολή είναι ανθρωπιστική. Είχαμε 10 συναντήσει, 70 ώρε συνομιλίε με του υπευθύνου και προσπαθούσαμε να βρούμε λύση. Δεν είναι μέρο του μνημονίου κατανόηση βεβαίω, αλλά στι 26 Δεκεμβρίου, μία μέρα μόλι μετά την υπογραφή και αφού θυσίασα τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου, πήγα στο Παρίσι για να συζητήσω το μνημόνιο συνεννόηση με τον κύριο Ρατζάβη και εννέα άλλου Είχα ακόμη άλλε εννέα συναντήσει κατά τη διάρκεια του 2012. Ναι, υπήρξε συμφωνία, δεν υπήρξε επίσημη υπογραφή, αλλά η διαδικασία εκκινήθηκε προκειμένου να σώσουμε τη ζωή των κατοίκων του καταπλησμού Και για να μην μπει ο στρατό του Ιράκ στον καταπλησμό. Εάν το έκαναν, πραγματικά θα γινόταν σφαγή διότι ο στρατό του Ιράκ ή η αστυνομία δεν μπορούν να ελέγξουν τα πράγματα. Είδαμε το επεισόδιο στη Χαβίντα πριν από δύο εβδομάδε, τρει περίπου εβδομάδε. Ο, ο σκοπό ήταν απλώ να ε, διαλυθεί μια διαδήλωση και 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του. Αυτέ είναι οι ανθρωπιστικέ αρμοδιότητε οι δικέ μου και των συναδέλφων μου. Σε ό,τι αφορά την παρέτηση. Α με ε, ενισχύσει και ο Γενικό Γραμματέα. Καλά είπατε βέβαια και εσεί και το απευθυνθήκατε και σα απήντησε. Ήταν σαφή η απάντηση, δόθηκε δημοσίω στο Συμβούλιο Ασφαλεία και στην τελευταία, με αφορμή την τελευταία έκθεση για το Ιράκ, στην παράγραφο 19, θα το θυμάστε. Το ξέρετε, εκφράστηκε εμπιστοσύνη και είπε ότι στηρίζει την προσέγγιση ω προ του καταβλισμού Άσραφ και Λίμπερτι και το πώ θα πρέπει οι άνθρωποι από, από αυτού του καταβλισμού να πάνε στο εξωτερικό. Υπάρχει αίτημα προ όλου που χρησιμοποιούν πόρους ε, ε, για τις ομάδες πίεση παγκοσμίω, αυτά τα χρήματα να τα πάρουν, να μην τα πετάνε στους ε, λομπίστε παγκοσμίω και να τα δώσουν στον καταβλισμό ΑΣΑΦ, Αυτή είναι η άποψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Μπανκιμούν. Επιτρέψτε μου να μην ζητήσω ποτέ παρέτηση. Πού το βρήκατε αυτό. Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του φυσικά. Αλλά εγώ θα μείνω και καλό θα ήταν να σκεφτείτε τι πολιτική συνεργασία μπορεί να υπάρχει αν από τη μια έχουμε την κυβέρνηση, από την άλλη την Αλκάιντα και από την άλλη του μουσουλμάνου αδερφού, του τους Σουφί, του Σουνίτε και ούτω καθεξή. Φυσικά δεν γίνονται όλα σωστά και δεν μπορεί να του ικανοποιήσει πάντα. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά όμω και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βεβαίω πάμε στου ανθρώπου και προσπαθούμε να συνεννοηθούμε. Φυσικά κάποιοι ζητάνε την παρατησή μου γιατί θεωρούν ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά μου. Αλλά τι να κάνω, να παρατηθώ. Αν παρατηθώ σε δύο μέρε στο Ιράκ, όλοι μπορούν να ζητήσουν την παρέτησή του. Αυτό δεν είχε γίνει στον καιρό του Χουσέιν, του Σαντάμ Χουσέιν. Κανείς δεν ζητούσε την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Σήμερα όλοι μπορούν να ζητήσουν την παρέτηση ενό Πρωθυπουργού, τη δική μου. Καλό είναι αυτό, δεν λέω. Είναι έκφραση ελευθερίας. Περιορισμένης μεν, αλλά ελευθερίας σε αυτή τη χώρα. Είναι πρωτόγνωρο για το Ιράκ αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπερβάλλεται σε ένα βαθμό. Έχω πολύ καλέ σχέσει με τον κύριο Λάουι και ποτέ δεν ζήτησα εγώ παρέτηση. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν θα ήθελα βέβαια να επεκταθώ σε αυτό. Απλά να σχολιάσω την παράγραφο 99 89 της εκθέση του Γενικού Γραμματέα που αφαίρεται και στις ε, ομάδε άσκηση πίεση ανά τον κόσμο και ζητά να ε, χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια και τα χρήματα που δοπανώνται εκεί για την επανεγκατάσταση, τη μετεγκατάσταση. Να σταθώ σε αυτά που είπαν κάποιοι βουλευτέ εδώ για τη μετεγκατάσταση και επαναπικεντρωθούμε σε αυτήν. Ειλικρινώ, δεν καταλαβαίνω πώ κάποιο λέει η ασφάλεια δεν είναι επαρκής στη χώρα, στον καταβλισμό Άσραφ και φυσικά καταδικάζονται τι τρομοκρατικέ επιθέσει τη 9 Φεβρουαρίου. Ήταν καταστροφικέ για όλη τη διαδικασία ερήρευση. Δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Όμω, ταυτόχρονα λένε, θέλουμε να μείνουμε στον καταβλισμό. Μα υπάρχουν 210, κύριε Χίγκινς, 210 άνθρωποι που μπορούν να πάνε στην Αλβανία και 100 στη Γερμανία. 310, έτσι είναι η σούμα. 310 έχουν προσφορές μεταγκατάστασης. Και εγώ ε, απευθύνθηκα σε εσά να ε, σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους πείτε να πάνε εκτός Ιράκ. Είναι επικίνδυνη η χώρα. Δεν τους συστήνω να μείνουν στο καταβλισμό Liberty. Και αν αποφασίσουν να μείνουν εκεί και να πούν ότι είναι αλληλέγγυοι, αλλά έχετε δίκιο. 14 όμω μόνο άτομα πήγαν στην Αλβανία μετά από 6 εβδομάδε. Εγώ το Φεβρουάριο συζητούσα με τον Περίσα και του υπεύθυνου τη ε, ΥΠΑΤΣ Αρμοστία για του πρόσφυγε του ΟΗΕ. Και προσπαθήσαμε να του πάμε από του 200 από. να διπλασιάσουμε τον αριθμό των ε, όσων θα μετεγκατασταθούν. Έχετε δίκιο. Είναι η μόνη διέξοδο αν είναι κακέ οι συνθήκε ασφάλεια. Αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια κανενό. Δεν είναι αρμοδιότητά μα, είναι αρμοδιότητα τη κυβέρνηση του Ιράκ αυτό. Στηρίζουμε του κατοίκου του Ασάφ ώστε να έχουν προστασία, να υπάρχει επιτήρηση. Αλλά η κυβέρνηση είναι ουσιαστικά ασφαλής για την προστασία. Είναι επικίνδυνος ο χώρος αυτός αναφέρθηκε ότι 700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες. Σας είπα, 85 έχασαν τη ζωή τους προχθές. 85 σκοτώθηκαν προχθές. Αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει να επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Γι' αυτό να φύγουν αυτοί από τη χώρα, να βρουν ασφαλές, ασφαλές καταφύγιο αλλού για την εκένωση, για την εκένωση να μας πείτε για την εκένωση. Με τρομάζει και εμένα αυτό ως γεγονός. Ωστόσο εδώ πρέπει να σας πω κάτι. Έχω φτάσει στο τέρμα των ικανοτήτων μου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο για τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε, τώρα για τα ονόματα των τριών δικηγόρων δεν έχουμε την ε, ε δυνατότητα να αναφερθούμε σε αυτό σε σχέση με τους τρεις δικηγόρους. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις τότε δηλαδή δεν θα ασκηθεί δίωξη από την κυβέρνηση για τις δραστηριότητες τους. Αυτό μας δόθηκε γραπτός. Το είπαμε πάνω από 10 φορές, πάνω από 12 φορές ότι θα έπρεπε να διοριστούν αυτοί οι δικηγόροι. Το Παρίσι δεν διορίζει αυτούς τους δικηγόρους. Εγώ ζητώ τη δική σας βοήθεια να τους πείτε αμέσως δώστε μας εμάς την άδεια να διαβιβαστούν τα στοιχεία αυτών των δικηγόρων Υπάρχει μια στενοπόσα αυτή τη στιγμή γιατί δεν απαντούν στα μηνύματά μας. Δεν μπορούμε όμως ε, να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε αν δεν είμαστε σε θέση να δράσουμε άμεσα. Εκένωση. σε σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη. Τι κάνει, τι κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη για την ασφάλεια. Εμείς ζητάμε πραγματικά κάθε εβδομάδα εκ νέου από την κυβέρνηση του Ιράκ να διασφαλίσει τις ε, οδηγίες και να βελτιώσει τους όρους ε, ασφάλειας. Ε, υπάρχουν 369 τέτοια καταλήματα και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα εκεί. Τώρα, σε σχέση με τα τυχώματα αυτά που αφαιρέθηκαν μετά από αίτημα των εγκατεστημένων εσείς εκεί, θα θυμόσαστε τη συζήτηση. Είπαν ότι είναι μια φυλακή. Πρέπει να αφαιρεθούν αυτά τα τυχώματα πρέπει να επιστρέψουν λένε κάποιοι. Ε, ποτέ δεν ε, είχα επέμβει στα θέματα ασφάλειας. Είχα όμως επιφυλάξεις για την αφαίρεση αυτών των τυχωμάτων που υπήρχαν εκεί όταν ήταν οι Αμερικανοί και για την ε, καταστροφή αυτών. Ποτέ δεν είπα ότι πρόκειται για ένα παράδεισο εκεί. Δεν είναι ένας χώρος στον οποίο θα ήθελα να ζω. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είναι προσωρινή αυτή η κατάσταση και να μπορούν οι εγκατεστημένοι στο Λίμπερτι να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και τελευταία παρατήρηση, πρόκειται για την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε αυτό το στρατόπεδο. Κάντε ό,τι περνάει από το χέρι σα να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση όσον αφορά τη διασφάλιση τη ελευθερία κινήσεων, τη ελευθερία πληροφόρηση, να μπορούν να μα μιλήσουν ελεύθερα, να μπορούν να συνεργαστούν ελεύθερα με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών και αφήνοντα την ιδιότητά μου των Ηνωμένων Εθνών στο περιθώριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τι αρχέ και αξίε των δικαιωμάτων του ανθρώπου και που ω Ευρωπαίο είμαι γι' αυτό, θα πρέπει τώρα εδώ να κάνουμε τι. Να αγνοήσουμε αυτές τις δομές στο στρατόπεδο Λίμπερτι όπου βρίσκονται σε τομείς ε, και ε, τμήματα και όπου υπάρχουν 30 καρτίνες αυτή τη στιγμή ώστε να μην επιτρέπεται να βρίσκονται σε, μία, σε ένα τέτοιο χώρο αυτοί οι άνθρωποι. Κλειδώνονται σε χώρους αυτοί, αυτά τα άτομα αν δεν επιθυμούν να έρχονται σε επαφή και να συζητούν με τους επόπτες μας. Αυτή είναι η σωστή πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τους Ευρωπαίους. Όχι, πιστεύω δεν είναι καθόλου σωστή. Και είναι υποχρέωση κοινοβουλευτικών εκπροσώπων να αντιμετωπίζουν όχι μόνο θέματα θανατικής ποινή και σωστό είναι αυτό να γίνεται και θέματα βασανιστήριων στις Ιρακινές φυλακές αλλά και να δούμε και τα θέματα υποστήριξης αυτών των δομών που όμως δεν δίνουν τη δυνατότητα ελευθερίας κινήσεων σε αυτούς τους ανθρώπους και την ελευθερία να εγκαταλείψουν αυτό το στρατόπεδο. Πρόσφατα κάποιο ε, έφυγε, χόλενε, έπεσε κάτω και τον τράβηξαν, τον έσυραν πίσω. Κανεί δεν παρενέβη. Και σε σχέση με την. Ε, ε, επιστροφή του σε αυτό το στρατόπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα επιτόπου και δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί αυτά τα γεγονότα τα αγνοούμε. Αγνοούνται σε μια οργάνωση η οποία έχει δεσμευτεί υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάντα έχει εγγράψει και εγγράφει τα δικαιώματα του ανθρώπου στην ημερήσια διάταξή τη και αυτό είναι σωστό, αλλά δεν πρέπει να αγνοούνται τέτοια γεγονότα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Κόμπλερ. Εχθές ε, με, μια, με ένα μήνυμα κάλεσα την κυρία Γιάννα Γνωσκόβα να έρθει στην Επιτροπή μας ώστε να ακούσουμε τα σε σχέση με την εξέλιξη, τις εξελίξεις στο Ιράκ και να προαγάγουμε τον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε σχέση και με την ε, δυνατότητα δηλαδή της ε, ε, πρόσκλησης στις Βρυξέλλες του υπευθύνου για τις, τα δικαιώματα του ανθρώπου του Ιρακινού Κοινοβουλίου. Νομίζω συνολικά οι δραματικές εξελίξεις καθίστανται ανάγλυφες θα πρέπει εδώ πραγματικά να φορά κανείς κράνη και να έχουν ε, γυλαίκα ε, που μπορούν να προστατέψουν από σφαίρες ε, τους κατόχους τους. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το να βρίσκεται κανείς εκεί. Και αν δει κανείς τις απειλές που διαμορφώνονται σήμερα εκεί, είχαμε, είπαμε τον ε, ε, Απρίλιο 750, 750 ε, θύματα. Δεν πρέπει εδώ να διαφοροποιούμε μεταξύ του ενός και του άλλου, πρέπει όλοι να προστατεύονται. Πρέπει φυσικά να βλέπουμε τι είναι δυνατόν, αλλά όμως υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες από τη διεθνή κοινότητα σε σχέση με σφάλματα που έγιναν ήδη κατά το παρελθόν. Ήμουνα πάντα κατά του πολέμου στο Ιράκ και είχα κρούσει κόδωνα κινδύνου για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράκ πριν από 10 χρόνια και είχα και προβλήματα και στη χώρα μου λόγω αυτής της θέσης μου. Όμως τα πράγματα έχουν ως έχουν και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτές τις επιπτώσεις, πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να πω τούτο, το ότι θα πρέπει να συζητήσουμε με τις χώρες μας, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εδώ έχουμε μεγάλη ανθρωπιστική πρωτοβουλία και δράσεις και δεν είμαστε σε θέση να διαθέσουμε από τις χώρες μας να υποβάλουμε προσφορές για να μπορούν να φύγουν από αυτά τα στρατόπεδα οι άνθρωποι αυτοί και να βρουν καταφύγιο στις χώρες μας. Η χώρα μου πάνω από 100, ε, περισσότερους η Αλβανία. Και τώρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε, ίσως είναι δυνατόν να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει αυτό. Πρέπει να δούμε και τα μεγέθη. Από ό,τι ακούω στο Camp Ashraf υπάρχουν 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα λέει. Στρούον. Και αν αυτό αληθεύει, δεν το ξέρω αν αληθεύει, γι' αυτό το εμβαδόν, πρόσφυγες που θεωρούνται παράνομοι στη Μεγάλη Βρετανία βρίσκονται σε ένα στρατόπεδο στο Σάσεξ με 30 λέει τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Σάσεξ ή στη δική μου χώρα. Ή... Ποια συζήτηση θέλουμε να έχουμε, ή στο Γκόλουε, ποια συζήτηση θα είχαμε στις χώρες μας αν είχαμε μια τέτοια κατάσταση σε αυτές τις περιοχές και βλέπουμε εδώ το θέμα του τριπλασιασμού ε, λόγω, αυτών των, ε, λόγω αυτής της κατάστασης. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και σωστοί. Λένε οι Ιρακινοί δεν τους θέλουμε αυτούς. Και ε, λέμε και εμείς ότι πολλές φορές δεν θέλουμε παράνομους μετανάστες στις χώρες μας. Και γι' αυτό είναι σκόπιμο να επομιστούμε τις ευθύνες μας και να μεριμνήσουμε αυτοί οι άνθρωποι να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε στις χώρες μας, στις πρωτεύουσές μας, να βρεθούν δυνατότητες για αυτούς. Αυτοί που έχουν επαφές σε σχέση με το ή το Cap Liberty, να βρουν μια δυνατότητα για αυτούς. Να υπάρξει δυνατότητα να φύγουν από το Ιράκ και να καταλήξουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ίσως προς όφελος των ανθρώπων εκεί. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε από κοινού αντί να, κάνουμε, να ε, κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, ώστε προς όφελος των ανθρώπων αυτών να λυθούν τα προβλήματά τους. Είναι απίστευτα αυτά που άκουσα σήμερα. Το διαδίκτυο να μην είναι λέει, διαθέσιμο με ελεύθερη πρόσβαση ατομική σε αυτούς τους ανθρώπους ή να μην υπάρχουν λέει, κινητά τηλέφωνα για αυτούς ή να υπάρχει μόνο ένας διά ένα κανάλι τηλεόρασης που εκπέμπει μόνο εκπομπές ε, προπαγανδιστικές. Δεν πιστεύω τα αυτιά μου, αλλά αν αυτά αληθεύουν έτσι έχω μεγάλο πρόβλημα, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό και θα ζητήσω να έχω πληροφορίες αν συμβαίνουν αυτά στο Καμπ Και εδώ σε σχέση όχι για παράδειγμα με την, τις απαιτήσεις των ΗΕ αλλά για την ηγεσία του στρατοπέδου αυτού κάτι να γίνει και σε σχέση με την τελική μου κρίση ε, φτάνουμε στο τελικό σημείο πρέπει να προσπαθήσουμε με αμερόληπτη τους αμερόληπτους οργανισμούς ε, να ενημερωθούμε σωστά ώστε σε αυτή τη συζήτηση να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια θέση να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Κόμπλερ για όλα όσα κάνατε σε αυτά τα δύο χρόνια που εσείς μέχρι σήμερα βρισκόσαστε στο Ιράκ υπό αυτή την ιδιότητα και εύχομαι αν δεν ξανασυναντηθούμε επίσημα για τη νέα σας αποστολή. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Και νομίζω με τη Γιάννα Ιβασκόβα θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να εξευρεθεί μια λύση σε αυτά τα προβλήματα. Φτάνει πια αυτό. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, να βοηθηθούν, να μας επιτρέψουν να τους βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πρόεδρος. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Θέλω να πω ότι είναι και κλεισμένο των θυρών θα εξεταστεί αυτό το σημείο. Παρακαλώ όσους δεν έχουν σχέση λοιπόν να εγκαταλείψουν την αίθουσα.